So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, let's continue. Our commissioner has arrived, so I... Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έχει έρθει ο Επίτροπος. Καλωσορίζω τον Επίτροπο κύριο Έρτιγκερ. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας ε, και μπορούμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σου για την δικασία απαλλαγής του 2017 και 2018. Να καλωσορίσω και το Γενικό Διευθυντή που είναι δίπλα σου και να σου δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Verehrte äh, Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, Σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας συναντήσω σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών. Και επειδή πολλοί από εσάς ε, βρίσκεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αλλά είσαστε καινούργοι και τα επόμενα πέντε χρόνια σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι Κατά κανόνα υπάρχει πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών και στην Επιτροπή Προεπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και με το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά ε, και με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν. Νομίζω αυτό το στοιχείο συμβάλλει στο ότι η δουλειά μας είναι αποτελεσματική, η Ευρώπη έχει προστιθέμενη αξία και αυτό που έχουμε κατορθώσει είναι να ε, είμαστε φιδωλοί στη διαχείριση των κονδυλίων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Αυτό βεβαίως το πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία από κοινού με τα κράτη-μέλη προβαίνει σε επενδύσεις. Ο Γενικός Διευθυντής Κραφ ε, προβαίνει στον εσωτερικό έλεγχο και αυτός ε, είναι πολύ σημαντικός πράγμα. Συμβάλλει προς την κατεύθυνση που σας παρουσίασα. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε το θέμα της ε, απόδοσης, των οικονομικών επιδόσεων μάλλον, να το προβάλλουμε να το προβάλλουμε προς τα έξω, τουλάχιστον κατά την τελευταία ε, θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς καλείστε να ελέγχετε το πώς εφαρμόζονται τα μέτρα. Ε, έχετε λάβει ε, εσείς ειδικά μέτρα και εμείς αυτά τα έχουμε θετήσει. Παραδείγματος χάρη θα ήθελα να αναφέρω την ανανέωση του κανονισμού που διέπει τον προπολογισμό τους ε, γενικότερους κανονισμούς, financial regulations. Αυτή είναι μια πολύ επίπονη εργασία, ήταν όμως πολύ σημαντική, κομβική σημασίας για να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο και να υπάρχει και ε, διαφανής ε, λογοδοσία να υπάρξει και απλούστευση πολλών διατάξεων. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, Έχουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. 160 δις είναι ο προπολογισμό αυτός. Τα τρία τέταρτα των κονδυλίων ε, διαχειρίζονται από τα κράτη-μέλη και ε, ταμιεύονται στους τελικούς χρήστες. Εμείς ε, επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από την ποιότητα της εργασίας, από τα Υπουργεία, από την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη και όλοι από κοινού καλούμεθα να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε οι κανόνες μας ε, να είναι κατανοητοί για όλους τους υπαλλήλους εκτός των Βρυξελών. Έχοντας λοιπόν κατά νου τα τελευταία τελευταία έτη επιτύχαμε πρόοδο. Επιτύχαμε καταρχήν το ελεγκτικό συνέδριο αντί να έχει κάθε χρόνο αρνητικό συμπέρασμα στην, στο τελικό του αποτέλεσμα, να αναφέρει ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει μία ουδετερότητα και υπάρχει σαφής ε, βελτίωση των θετικών αποτελεσμάτων. Τα τελευταία χρόνια μειώθηκε ουσιαστικά το, το, ποσοστό σφάλματος, έχει φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο και ε, εδώ και χρόνια η αιτήση, η υπολογισμοί και οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κρίνονται ως ε, ικανοποιητικοί. Υπάρχει καλύτερη καταπολέμηση της απάτης. Ε, έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος για να ε, επιτευχθεί η καταπολέμηση της απάτης. Η Όλαφ ε, είναι ανεξάρτητη, είναι αποτελεσματική, είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής εισαγγελία ε, στον αγώνα για την καταπολέμηση της απάτης και η Όλαφ είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω σήμερα να εγκρίνετε τον κανονισμό που διέπει την Όλαφ, ο οποίος ανανεώνεται και το αργότερο μέχρι του τέλος του έτου θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναλάβει τις εργασίες της. Εσείς έχετε επιτύχει να μπορείτε και να έχετε λόγο στην εκλογή ε, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Στο μέλλον θα υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην ε, Όλαφ και τον ε, Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, όπως ορίζει το άρθρο 883. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και την έννοια ενός μιας δέσμης ε, από ε, απολογισμούς. Αυτό είναι ένα κομμάτι του κανονισμού ε, του προϋπολογισμού. Πέντε τμήματα περιλαμβάνει αυτή η δέσμη των ε, ε, ισολογιστών εκθέσεων. Καταρχήν έχουμε τα αιτήσια μέτρα, μέτρα τα οποία προβλέπονται για την απαλλαγή του προηγούμενου έτους. Εδώ μιλάμε για το 2017. Μετά είναι η έκθεση για τους εσωτερικούς ελέγχους την περασμένη χρονιά. Για πρώτη φορά θα κατατεθούν μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και για τη δομή του. Στη δέσμη αυτή για κάθε ευρώ αναφέρεται πώς δαπανήθηκε αυτό το ευρώ και το τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε η διοίκηση να ανέβει στο ανώτατο επίπεδο. Στη δέσμη αυτή ε, συζητήσατε, ε, πρόσφατα τοποθετηθήκατε και εγώ θα ήθελα τώρα να εστιάσω την προσοχή μου στην, ε, στο βασικό νόημα αυτών των εκθέσεων. Η ετήσια, ο ετήσιος απολογισμός διαχείρισης και οικονομικών επιδόσεων. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη για τη διαχείριση του προπολογισμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση για την περασμένη χρονιά. Με αυτόν τον απολογισμό προκύπτει μια γενική εικόνα για τους στόχους αλλά και για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. Δίδουμε πληροφορίες για τα αποτελέσματα που επιδιώκει ο προπολογισμό με βάση τι πολιτικές και τα προγράμματα. Πέρυσι λοιπόν είχαμε στον προπολογισμό μα δύο προτεραιότητε. Πρώτον, την υποστήριξη τη οικονομική κατάσταση, τη σταθεροποίηση της οικονομία και τη αγορά εργασία και δεύτερον, την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, συγκεκριμένα, ε, κλασικά παραδείγματα και χειροπιαστά παραδείγματα για αυτά που σας είπα. Από το 2015 μέχρι πέρυσι, με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ακτοφύλακης, κατορθώσαμε να συμβάλλουμε στην διάσωση 690.000 ανθρώπων ε, στη θάλασσα θα θυμάστε πολλές ε, τρομακτικές εικόνες, ε, νεκρούς, ε, πνιγμένους, αλλά εμείς με τα ευρωπαϊκά μας μέτρα κατορθώσαμε να κάνουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεύτερον, με το εργαλείο των προσφύγων και της Τουρκίας κατορθώσαμε ε, να κατασκευάσουμε περίπου 150 σχολεία, ε, να δώσουμε δυνατότητα πάρα πολλά παιδιά να επισκέψουν το σχολείο. 60.000 ε, παιδιά μπόρεσαν να χωρίσουν τις σπουδές τους. Έχουμε τώρα περίπου 650.000 παιδιά προσφύγων τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Αυτό είναι η ελάχιστη προσφορά μας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην παιδεία για να υπάρχει προοπτική. Πέρυσι για 800.000 δασκάλους ε, και ε, βοηθούς δασκάλων ε, στο εξωτερικό δώσαμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Ή στην έρευνα μπορέσαμε να εφαρμόσουμε την πρωτοβουλία μας για την κβαντική τεχνολογία. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς ερευνητές και με τον τρόπο αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, κυρίως στον τομέα της κβαντοτεχνολογίας. Επιπλέον, κατορθώσαμε να στηρίξουμε και να εφαρμόσουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσφατα προσπαθήσαμε με το Discover EU να ε, δώσουμε τη δυνατότητα σε 15.000 ανθρώπους ε, να ταξιδέψουν στην Ευρώπη με το τρένο δωρεάν. Και ε, στην ε, αντιμετώπιση καταστροφών, στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. Επτά αεροπλάνα, έξι, ε, έξι ελικόπτερα χρηματοδοτήθηκαν και οργανώθηκαν από εμάς. Επιπλέον, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο του 20%, το 20,7 των δαπανών μας ε, διοχετεύτηκε στην προστασία του κλίματος, στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου ε, του άνθρακα, εκπομπών θερμοκηπίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι η εσωτερική διαχείριση του προϋπολογισμού και γι' αυτό σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη εφαρμόσαμε συστήματα ελέγχου έτσι ώστε όλες τις δαπάνες να τις καταστήσουμε συμβατές με τους κανόνες. Η καταβολή σε αδυνάμους ε, χρημάτων που δικαιούνται χωρίς ε, καμία καθυστέρηση και χωρίς ε, γραφειοκρατικά προσκόμματα. Επίσης, στην περίπτωση που εντοπίστηκαν αχρεωστήτως καταβλητέντα, ανεκλήθησαν τα ποσά αυτά. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει και διαφάνεια για ε, αδυναμίες, αδυναμίες ε, για τις οποίες προσπαθούμε να λάβουμε διορθωτικά μέτρα. Εξάλλου μας ενδιαφέρει και η πρόληψη στο μέλλον ε, να μην γίνονται τα ίδια λάθη, να αποφεύγονται τα λάθη αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι με όλα τα μέτρα αυτά μπορούμε να διεκδικήσουμε την υποστήριξή σας in-camera control. Αυτό είναι έλεγχος όσων εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η δεύτερη προτεραιότητά μας. Ε, τα συστήματα αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Μπορέσαμε να επιτύχουμε μετά την εφαρμογή όλων των ελέγχων ε, το, ποσό, το ποσοστό όσων παραμένουν να είναι κάτω από το 2%. Πέρυσι υπολογίζουμε ότι το ποσοστό αυτό είναι στο περίπου 1%. Ε, Πέρυσι επίσης ε, προβήκαμε σε ε, διορθώσεις που ανέρχονται σε περίπου 6 δις ευρώ. Αυτό αφορά το προηγούμενο έτος και τα έτη αυτού. Τα χρήματα θα διοχετευτούν στον κανονικό προϋπολογισμό. Οι αιτήσιοι λογαριασμοί μας είναι ο κρογονέος λίθος του, της έκθεσής μας, γιατί θέλουμε να έχουμε μια περιεκτική, διαφανής εικόνα όλων των χρηματοπιστωτικών στοιχείων, τόσο όσον αφορά τα έσοδα, όσο και στα έξοδα. Το ελεγκτικό συνέδριο για το 2017 κατέληξε σε θετικό συμπέρασμα, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Στις 8 Οκτωβρίου θα καταθέσει σε εσά άμεσα το συμπέρασμά του. Είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει. Ε, διάκυμε ε, αισιόδοξο, συγκρατημένα αισιόδοξο. Και επειδή μας παρακαλέσατε θα συνεχίσουμε και φέτος ε, τον, την έκθεσή μας να την καταθέσουμε ένα μήνα νωρίτερα έτσι ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία της απαλλαγής να ολοκληρώνεται νωρίτερα. Ας δούμε τώρα λιγάκι ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές μας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εφέτος για πρώτη φορά ε, θα καταθέσουμε μία μακροπρόθεσμη προοπτική, όπως ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους ετήσιους υπολογισμούς θα συμπληρωθούν με προβλέψεις για τα επόμενα πέντε έτη. Σήμερα λοιπόν η έκθεση καλύπτει την περίοδο 20 μέχρι 24 αυτό που μας ενδιαφέρει υπάρχει ένα σχέδιο για το πλαίσιο που όμως δεν έχει ακόμα εγκριθεί και με βάση αυτό το σχέδιο θα έχουμε τις προβλέψεις μας, δαπάνες, μάλλον έσοδα, έξοδα, αυτά μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής της θητείας. Όσον αφορά τώρα τα προσεκαθάριση ποσά, θα Θέλω να πω επ' αυτού ότι αυτά τα προσεκαθάριση ποσά, τα ραλ, είναι κατ' ουσίαν ε, το άθροισμα των ε, υποχρεώσεων που δεν έχουν γίνει ακόμα πληρωμές. Το θέμα που τίθεται είναι πότε ακριβώς ε, θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι υπολογισμοί τους έτσι ώστε να μπορούν να καταβληθούν τα ποσά. Γιατί τα ποσά θα καταβληθούν και όσο το νωρίτερα τόσο καλύτερα. Όμως ε, είναι ξεκαθαρισμένο το θέμα ε, των ε, πληρωμών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην καταφτάσουν όλοι οι υπολογισμοί μαζί, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα για το μέλλον και να μπορέσουμε να επιτύχουμε την έγκριση του Συμβουλίου. Με την δέσμη τη δική μας, ε, βεβαίως και ικανοποιούμε σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματά σας. Παραδείγματο χάρη, όσον αφορά την έκθεση για τα μέτρα που θα ακολουθήσουν Θέλω να πω επ' αυτού τα εξή. Πρώτον, όσον αφορά την επίδοση, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει ε, μια ανανέωση του προπολογισμού για το επόμενο πλαίσιο. Προτείνουμε σημαντικέ αλλαγέ. Επίση, ε, καθορισμό σαφών στόχων ή αν θέλετε Εκεί θα υπάρχουν μικρότεροι δείκτες ε, υψηλών οικονομικών επιδόσεων. Όσον αφορά στον διορισμό ε, ανώτερων υπαλλήλων, ε, και εμείς μόνοι μας εξετάσαμε το ποιες ήταν οι διαδικασίες μέσα στην ίδια την Επιτροπή. Αυτό που θέλουμε να εφαρμόσουμε είναι το STEP Regulation και να δούμε και ποιες είναι οι ειδικές σας απαιτήσει έναντι ημών. τον καιρό που μου απομένει μέχρι να ολοκληρώσω τη θητεία μου θα καταθέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ε, προτάσεις μου με βάση την εμπειρία μου για να υπάρξει βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Περνάμε τώρα στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σας ενημέρωσα πολύ συγκεκριμένα για μέτρα που ελήφθησαν για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου η εφαρμογή αυτή ελέγχθηκε μέσα από ελέγχους, μέσα από audits και ελέγχθηκε το κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί. Επ' αυτού θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με διαφάνεια, κυρίως έναντι ημών. Αποφασίσαμε, παραδείγματο χάρη, ότι ε, Όσον αφορά τις συστάσεις ε, του διαμεσολαβητή για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα, αυτό ε, στο βαθμό του δυνατού θα μπορέσουμε να το ικανοποιήσουμε. Και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενημερώσω το Κοινοβούλιο επ' αυτού και θα σας παρακαλέσω βέβαια να διαφυλάξετε και την απαραίτητη εχεμήθεια θα σας ενημερώσουμε για τους ελέγχους που έγιναν, που διεξήχθησαν πέρυσι. Ο ε, Γενικός μας Διευθυντής, ο κύριος Κραφ, που είναι και σήμερα παρόν, είναι και συνομιλητής σας, είναι εκείνο που έκανε τους ελέγχους αυτούς. Με την εργασία της δικής του της ομάδας ε, διαφυλάσσουμε ε, την ε, εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εκτελεστικούς οργανισμούς. Οι δική του λοιπόν οι έλεγχοι θα οδηγήσουν βεβαίως και σε βελτίωση στο μέλλον. Για την περασμένη χρονιά έχουμε την έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή, ο οποίος καταλήγει στο ότι τα εσωτερικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολό τους λειτουργούν, παρότι βέβαια μεμονωμένα υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Αυτές τις αδυναμίες ε, τις αντιμετωπίζουμε, γι' αυτό το λόγο ο μεγάλος αριθμός των συστάσεων που εφαρμόστηκαν είναι η βάση τη μελλοντική μας εργασίας. Τελειώνω λοιπόν. Πρόκειται για την προστιθέμενη αξία. Προστιθέμενη αξία που ε, δημιουργεί ένας ε, προϋπολογισμός, ε, πρόκειται για προτεραιότητες. Νομίζω ότι όσον αφορά τον προϋπολογισμό μπορούμε να δείξουμε στον πολίτη ότι πραγματικά έχει νόημα να επενδύει κανείς ευρωπαϊκά. Και εδώ θέλω να παρουσιάσω τρία βασικά προβλήματα πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Πρώτον, η έγκαιρη έγκριση του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή είναι απόλυτη προϋπόθεση για να εφαρμόζεται ο προεπλογισμό ήδη από τον Ιανουάριο. Είμαστε στο 12 παρα 5 και θέλω να σας πω υπάρχουν ε, ε, απαιτήσει έναντι των ε, αρχών του προεπλογισμού υπάρχουν και εναντί του Συμβουλίου και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να κρίνουν και αυτοί ότι η έγκριση του προπολογισμού μέχρι το 27 είναι και για αυτούς πρώτη προτεραιότητα. Μετά ε, να ξεκινήσουν στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων τομεακές προτάσεις και να καταλήξουν σε συγκεκριμένους αριθμούς. Να δείξουν προτιμία ε, για συνδιαλλαγή το νέο κοινοβούλιο ε, πρέπει να έχει αυτή τη διάθεση τη συνδιαλλαγή. Ορισμένα κράτη-μέλη βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ πρόθυμα. Όσον αφορά στα κράτη-μέλη και τις αρχές, εθνικές και τοπικές αρχές, εξαρτώμεθα από αυτές και για το λόγο αυτό ε, και σε αυτό το επίπεδο και όχι απαραίτητα στο επίπεδο της Επιτροπής πρέπει να υπάρχει μια βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Έχουμε την ε, πολιτική συνοχής η οποία καλείται να εφαρμόσει 390 προγράμματα ε, στις περιφέρειές μας. Στον τομέα της ε, συνοχής, κράτη που γίνονται στα κράτη-μέλη, προφανώς και μετακυλίονται, έχουν επιπτώσεις σε εμάς. Στον τομέα δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακών Υποθέσεων και Απασχόλησης μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ένας πολύ σημαντικός μας εταίρος. Έχουμε κοινά ε, σημεία αναφοράς. Το ελεγκτικό συνέδριο μας παρακολουθεί, μας συνοδεύει και εμείς στηρίζουμε το ελεγκτικό συνέδριο. Αν, θα το στηρίξουμε αν θα θελήσεις να ε, αναθεωρήσει τους ε, κανονισμούς. Και τέλος πρέπει όλοι από κοινού να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι βασικότεροι παράγοντες για την μέτρηση ε, της απόδοσης και για την προστιθέμενη αξία αυτά να κρίνονται με τέτοια κριτήρια. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να ε, κρίνει και να αξιολογήσει κανείς τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά νομίζω ότι επ' αυτού επιτύχαμε αρκετά. Ε, καθαρά μηχανική μέτρηση, αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Να περάσουμε σε πιο ρεαλιστικούς ορισμούς για το τι ακριβώς είναι η οικονομική επίδοση. Υπάρχει η διαδικασία απαλλαγής για πέρυσι που αφορά την Επιτροπή Juncker και κατά τους πρώτους μήνες της επόμενης Επιτροπής, τότε θα υπάρξει η απαλλαγή. Ε, αν πρόκειται να θυγεί ο παλιός προϋπολογισμός, ε, νομίζω ότι τότε θα πρέπει να εξεταστεί στην δική σας την Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν θα υπάρχει αυτή η μεταβατική φάση που πρέπει όλοι από κοινού να την περάσουμε ικανοποιητικά και παρόλα αυτά να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε, έχω την τιμή να είμαι εισηγήτρια για την απαλλαγή των προεπλογισμών του 2018, οπότε θα μου τρέψετε να ξεκινήσω εγώ το γύρο των ερωτήσεων αν και ίσως να μην είναι απόλυτα σωστό, τέλος πάντων ε, θα ξεκινήσω εγώ ως εισηγήτρια. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις ε, προς εσάς. Πρώτα απ' όλα, είπατε ότι πολλά έχουν επιτευχθεί ε, και εδώ έχω μια ερώτηση σε σχέση με την αναφορά των επιδόσεων, διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις για το τι θα πει αυτή η αναφορά επιδόσεων και τελικά ε, και θέλει κανείς ε, να προωθήσει ε, στοιχεία τα οποία να είναι εύληπτα, διαφανή και να δείξει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Όμως τελικά υπάρχουν αντιφάσεις και αδιαφάνεια. Το ΡΑΛ, το υπόλοιπο προσεκαθάριση. Ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι στη ΓΔΡΕΓΙΟ... ΡΕΓΙΟ... Εκεί ε, υπάρχουν καθυστερήσεις ε, λόγω του κανόνα συντρία ε, και η γάμα δέλτα Ρέγγιο πιστεύει μαζί και με τη δική μας την πρέπει να πάει λίγο πιο γρήγορα το πράγμα. Η ερώτηση μου είναι για το επόμενο πολιετές από πλευρά της Κομισιόν θα πάτε στο νησιν 2 μήπως γιατί ο κανόνας του νησιν 3 αποτέλεσμα πάνω από το 50% των πληρωμών να, να γίνεται στο επόμενο πολιετές και αυτό δεν διευκολύνει και τόσο το έργο για την επεξεργασία ενός νέου πολιετούς, ε, ιδίως με βάση τις ε, απαιτήσει και τους όρους που υπάρχουν. Επόμενο ερώτημα. 0,8% ε, μόνο είναι το ποσοστό σφάλματος. Με εκπλήσει αυτό και με εντυπωσιάζει. Πώς είναι δυνατόν 0,8% Είχαμε τη συζήτηση και με την Επιτροπή και με το ελεγκτικό ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία σε σχέση με τα στοιχεία που δίνουν οι δύο. Ε, μετά από τις διορθώσεις διαφορετικά τα ποσοστά. Η Κομισιόν λέει ότι εμείς κάνουμε πράγματι κάποιες διορθώσεις ε, Θέλουμε να λειτουργούν σωστά και λειτουργούν σωστά οι έλεγχοι, αλλά πράγματι ε, είναι πιο ψηλό το ποσοστό πριν τις διορθώσεις και αυτό είναι ένα δείγμα που δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα ε, με την εκτέλεση των προγραμμάτων. Γι' αυτό και το ερώτημά μου είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και πού ε, οφείλεται το σφάλμα σε κάθε περίπτωση, ποιες είναι οι πηγές των σφαλμάτων, ε, πρέπει να γίνονται διορθώσεις, ε, γιατί δεν θέλω να ασκήσω κριτική βέβαια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλό είναι να ανακαλύπτουμε και να διορθώνουμε τα πράγματα, της αδυναμίας, αυτό είναι σίγουρα θετικό, όμως παρόλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί χάνονται χρήματα. Ε, τα οποία θα πρέπει να εκταμευθούν, να καταβληθούν και ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία επιστρέφουν στις τσέπες των κρατών και δεν γίνεται και μια δίκαιη ανακατανομή δυστυχώς περισσότερες περιπτώσεις. ενώ θα χρησιμοποιούνταν καλύτερα στο πλαίσιο του νησιακού προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, πράγματι είναι και ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον μα για το θέμα αυτό. Σε ποιο βαθμό έχουμε κάποια αποτελέσματα για Σλοβακία, Τσεχία, είχαμε κάποια ζητήματα και με τη Ρουμανία ανέκυψε ζήτημα, Πολωνία επίσης. Ε, ίσως θα ήταν δυνατό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ε, σε ένα τρόπο ε, διαχείριση που θα μας δίνει περισσότερη ενημέρωση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο άτομο, με ενδιαφέρει πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με ενδιαφέρει τα βασικά και δεν με ενδιαφέρει τι θα ασχοληθεί μετά η δικαιοσύνη και οι ελεγκτικές αρχές. Ε, μόνο ίσως ε, εάν ε, είναι κάποιο εξέχον πρόσωπο. Εγώ πάντως γενικώς επιφυλάσσομαι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κάποιος προβεβλημένος ή όχι. Με ενδιαφέρει η δομή που κρύβεται από πίσω. Αυτές ήταν οι δικές μου ερωτήσεις και τώρα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στην κυρία Πένκοβα. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε για την παρουσία σας. Δύο ερωτήσεις έχω, σύντομες. Η πρώτη συνδέεται με το ερώτημα το οποίο έθεσε ήδη η κυρία Χολμάγερ αναφέρεται στη διαφορά της ορολογίας στα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι διαφορετικές γενικές διευθύνσεις και στην ε, ετήσια έκθεση επιδόσεων. Κατανοείτε αυτό το οποίο εννοώ. Μπορείτε να μας δώσετε εξηγήσεις λοιπόν τις διαφορές, για τις διαφορές, στην ορολογία την οποία χρησιμοποιούν οι διαφορετικές ε, υπηρεσίες οι γενικές διευθύνσεις. Είναι δύσκολο να συγκρίνει κανείς τα ποσοστά λάθους ε, και να καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα. Ε, και δεύτερον, αναθεωρημένες προβλέψεις για τις αυξημένες καθυστερημένες ε, πληρωμές για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί βλέποντας το πώς έχει εξελιχθεί ε, στις πιστώσεις υποχρεώσεων το τρέχον ε, πολιετές δημοσιονομικό. Και για την έκθεση follow-up ε, για το 2018 λέγεται ότι για δεύτερη χρονιά δεν χρειάστηκε ε, διορθωτικός προϋπολογισμός για τα τα ταμεία. Ε, πόσο μπορείτε να μας σχολιάσετε αυτή τη συγκεκριμένη φράση από την έκθεση follow-up. Ολιβιέ ή η Μαρτίνα μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για όλα κύριε Έτιγκερ. Έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια για θέματα απαλλαγής, ελπίζω να μην σας επιβαρύνουμε και ελπίζω να πάνε όλα καλά για σας και να μας λείψετε. Ή να σας λείψουμε εμείς μάλλον. Έχω και εγώ έχω κάποια ερωτήσεις σε σχέση με τα ποσοστα, ποσοστά λάθους και θα ήθελα να μάθω για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελεγκτικό συνέδριο σε επίπεδο ε, προσμέτρησης ποσοστών λαθών. Ε, εμείς ζητήσαμε να υπάρξει μια εναρμόνιση στη μεθοδολογία. Η Επιτροπή είπε ότι χρησιμοποιεί μια ενιοποιημένη μορφή αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις διαφορές που υπάρχουν ε, ανάμεσα στα διαφορετικά πεδία. Αυτό σημαίνει ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν ανταποκρίνεται στα ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ε, τι μπορούμε να ζητήσουμε από το ελεγκτικό συνέδριο, να ταυτιστεί με την ε, εναρμόνιση στην οποία προχώρησε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία τα σχετικά με το 18 χωρίς τις τελικές διορθώσεις θα είναι αντίστοιχα με τα στοιχεία του ελεγκτικού συνεδρίου. Και δεύτερον, τι γίνεται ακριβώς με την εξέταση των ε, συνδέσμων ανάμεσα σε δύο πλαίσια, στόχοι από τη μία και δείκτες από την άλλη, στον τομέα των επιδόσεων του προϋπολογισμού. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για το επόμενο στρατηγικό και προγραμματικό κύκλο. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταλήξουμε σε καλύτερα συμπεράσματα, σταθμίζοντας από τη μία τους δείκτες επιδόσεων και από την άλλη την επίτευξη των στόχων. Κοιτάξτε, είμαστε τελικά ιδιαίτερα τεχνικοί σε κάποια θέματα στην Επιτροπή αυτή αλλά έχουμε κάνει δουλειά και έχετε κάνει και εσείς δουλειά, έχουμε εργαστεί μαζί εσείς, το γραφείο σας και η Γενική Διεύθυνση Μπάντζου. σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκθεσή σας κύριε Επίτροπε. Ε, εγώ ε, δεν είχα μέχρι σήμερα την ε, χαρά να σας υποβάλω ε, ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας, αυτή που ακούσαμε σήμερα. Μεταξύ άλλων, είπατε, αναφέρατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το γεγονός ότι εγκρίθηκε αυτό. Βεβαίως και ε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτοβουλία της Επιτροπής. Βέβαια, η θέση του Προέδρου δεν αρκεί και νομίζω ότι είναι προς όφελος όλων μας το να είναι σωστά ε, ε, επανδρομένη η αυτή η Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πρόταση Επιτροπής, ε, γιατί αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την απάτη, χρειαζόμαστε πολύ καλή σύνθεση της Ευρωπαϊκής Συγγελίας, κάτι το οποίο δεν συμμερίζονται όλα τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο που μας απασχολεί αφορά βέβαια στις, ε, στα κονδύλια, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί το 2017. Νομίζω ε, είναι περίπου στα 260 δις και υπάρχουν και τα άλλα 150 δις που προκύπτουν συνήθως. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να ρωτήσω τελικά ε, πώς θα, πώς θα αντιμετωπιστούν, πώς θα τα διαχειριστείτε αυτά τα ποσά. Και τέλος, ε, θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να μην το κατάλαβα καλά, είπατε ότι θα υπάρχουν λιγότεροι δείκτες, αλλά εγώ από κάποια σχέδια είδα ότι σε πάρα πολλά θέματα ζητάτε περισσότερα στοιχεία και για την αξιολόγηση θα χρησιμοποιούνται περισσότεροι δείκτες. Και αυτό σημαίνει ότι για πολλούς οι οποίοι ασχολούνται με τις αιτήσει, ε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ε, υπάρχει μεγάλη απλούστευση κατά την εφαρμογή. Ίσως να μην το κατάλαβα καλά, ίσως ε, θα μπορούσατε λιγάκι να το διευκρινίσετε. Όλα τα άλλα έχουν ήδη υποθεί. Η Κορίνα. Uh, thank you very much, dear. Σας ευχαριστώ πολύ ε, Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είστε μαζί μας γιατί η απαλλαγή για το 2017 ήταν κάτι το σημαντικό. Νέες προκλήσεις εμφανίστηκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι κάνατε τα δύνατα δυνατά έτσι ώστε να μπορέσετε να συμπεριλάβετε θέματα όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, Frontex, άμυνα. Έχουμε ξεκινήσει και αρκετές αλλαγές στα λειτουργικά προγράμματα. Υπάρχει το παράδειγμα της Σουηδίας, αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν αλλάξει για να τα καταστήσουμε ε, ικανά να αγοράσουμε σκάφη για να σώσουμε ζωές στη Μεσόγειο και σας ευχαριστώ για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Η ερώτησή μου αναφέρεται το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό. Είπατε ότι είναι, είμαστε στο παραπέντε και πράγματι έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα και ακριβώς γι' αυτό ανησυχώ ε, αν δεν γίνει δεκτό το πολιετές μέχρι το τέλος του χρόνου, τότε η Ευρώπη θα βρει μπροστά της πάρα πολλές δυσκολίες γιατί εκατομμύρια φοιτητών δεν θα ωφεληθούν από το Εράσμους και από το Horizon 2020. Φυσικά εγώ μιλώ σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να είμαι δίκαιη και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε καλά τη δουλειά της και ξεκίνησε τις συζητήσεις από το Μάιο του 18, ενώ τώρα είμαστε στον Οκτώβριο. Ε, πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει μια κοινή προσπάθεια ανάμεσα στην Επιτροπή και στο ε, Κοινοβούλιο έτσι ώστε να πιέσουμε το Συμβούλιο επιτέλους να υιοθετήσει το πρόγραμμά του. Η τελευταία μου ερώτηση αναφέρεται τον Brexit. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει 15% μείον στον προϋπολογισμό. Αλλά συνολικά υπάρχουν, ε, προβλέπονται μειώσεις σε πολλές πολιτικές πολύ υψηλότερες. Δεν ξέρω τι, τι άποψη έχετε εσείς ε, ως πολιτικός, όχι μόνο ως επίτροπος. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία το Brexit ε, θα γίνει με άτακτο τρόπο. Το βάρος ε, δεν θα πέσει σε εμά στις Βρυξέλλες, θα πέσει στα κράτη-μέλη και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Μου και Κούς και μετά ο Επίτροπος γιατί έχετε ολόκληρο... Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις, απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για το International Management Group εάν δεν τηρηθούν αυτά που ζητάμε στις 26 Μαρτίου ε, με ψήφισμά μας, ούτε τηρηθούν αυτά που λέει η ε, δικαιοσύνη. Αυτό το EMG, το ΜΚΟ σε εμπόλεμες ζώνες, έχει εργαστεί αποτελεσματικά σε πολύπλοκες καταστάσεις, σε, σε περιοχές που πλήττονται από εμπόλεμη σύραξη κτλ. Γιατί έχετε τέτοια ε, προβλήματα και κάνετε τέτοια επίθεση σε, αυτό το, σε αυτή τη ΜΚΟ εδώ και χρόνια που έχει 200 άτομα που ενδεχομένως να χάσουν και τη δουλειά τους. Δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε. Γιατί τέτοιο κόλλημα και γιατί τέτοια έλλειψη διαλόγου. Γιατί επιλέξατε τη διαμάχη την ε, δικαστική και όχι το διάλογο. Γιατί δεν κάθεστε στο τραπέζι με εκπροσώπους του MG για την αναζήτηση μια, ενός φιλικού διακανονισμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χολμάιερ, και η ε, την Έχω υπηρετήσει ως ε, ερετός, ω δημοσιοπάλληλος στο Δήμο της Βάσης Βεργέρης. Έχω μια ερώτηση. Είστε Επίτροπος αρμόδιος ε, όχι μόνο για τον προϋπολογισμό, αλλά ξέρετε και για το προσωπικό της ε, περικοπές προσωπικού ε, και τι προβλήματα δημιουργούνται. Στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προβλέψεων υπάρχουν κάποια σχέδια να περιοριστεί το κόστος προσωπικού και αν ναι, τι σχέδια υπάρχουν. Γιατί το λέω αυτό. Διότι είναι ένα πρόβλημα και ε, ε, ασκούν κριτική όχι μόνο οι ευρωσκεπτικιστές αλλά και άλλοι για αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι είναι πολύ ψηλό το κόστος του προσωπικού και η μισθή, ιδίω ε, των διοικητικών υπαλλήλων, είναι πολύ ψηλή. Lieber Herr Kommissar, Frau Vorsitzende, äh, Damen und Herren, Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές, καταρχήν όσον αφορά το performance reporting, ε, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να επιδιώκουμε την εναρμόνιση των διαφόρων προγραμμάτων και των διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουμε αυτή την εναρμόνιση. Ας πούμε, στο Erasmus Plus, εκεί αναφέρεται πόσοι άνθρωποι κάθε χρόνο που πήγαν, ποτέ έφυγαν, ποτέ ήρθαν. Κανονικά αυτά είναι προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται μέσα σε ένα χρόνο στο Rail Baltica Εκεί ε, υπάρχουν ε, δεκαετή προγράμματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο το ε, να βρει κανείς συγκρίσιμα παραδείγματα ανάμεσα στο Connecting Europe, τη μετανάστευση, το Erasmus Plus. Ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχουν τεράστιες διαφορές, διαφορετικοί κόσμοι. Γι' αυτό λοιπόν παρόλα αυτά πρέπει να εναρμονίσουμε ε, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα πλαίσιο για να είναι δυνατόν να κατατίθενται και εκθέσεις. Σε γενικές τώρα γραμμές, ε, στη Βάδη Βιτεμβέργη, ένας προπλογισμός κρατηδίου ή αν θέλετε ας πάρουμε ένα κράτος όπως είναι η Βουλγαρία. Είναι ένας ε, προπλογισμός διαχείρισης που αφορά τους ε, ε, δασκάλους, ε, όλο τους υπαλλήλους. Μέχρι το 60% είναι ο προπολογισμό αυτός. Σε εμά όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η διοίκηση που αντί εκεί είναι 60% σε εμά είναι 7%. Και το 8% περίπου τόσο αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά έχουμε το 7% που είναι κομισιόν, κοινοβούλιο, στο οποίο παρεμπιπτόντως τώρα θέλουμε να δώσουμε ως μόνο θεσμό και νέες οργανικές θέσεις το ε, Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ε, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, 20.000 παιδιά. Αυτά περιλαμβάνονται στο δικό μας τον προϋπολογισμό. Νομίζω λοιπόν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε κάνει περικοπές. Αυτά φαίνονται από τους προϋπολογισμούς. Κοιτάξτε, μόνο ο Δήμος του Μονάχου έχει περισσότερους υπαλλήλου από την Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργοί από τα κρατήδια έρχονται εδώ με μία συνοδεία 10 ανθρώπων. Για δέστε, εγώ έναν έφερα. Και ξέρω, α πούμε, κάποια δημοτικά συμβούλια ε, στη Βαδβιτεμπέργη, αλλά και αλλού, αλλά και στην Αυστρία. Ε, και εσείς από την Αυστρία ε, πολυπληθήσει η παρουσία σας οποτεδήποτε φεύγετε από το Ζάλτσπρουκ, το Ινσπρουκ, τη Βιέννη και έρχεστε εδώ. Ή ε, σε νέα κρατήδια έρχονται πάρα πολλοί σύνοδοι. Σχεδόν τώρα θα έχουμε ανακάτοικο και υπουργό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί λόγοι που οδηγούν στο ότι ο ε, φορολογόμενος θέλει περικοπές. Το πετύχαμε αυτό. Το πετύχαμε εμείς αυτό. Όσον αφορά τους μισθούς. Και ναι και όχι θα πω εδώ από το 2014 κάναμε πολλά. Για δύο χρόνια πάγωμα, μετά μικρότερες αυξήσεις, αυξήθηκε ο χρόνος εργασίας, το ωράριο εργασίας. Σήμερα διαπιστώνω ότι από τα κράτη-μέλη κανείς δεν θέλει να έρθει στις ε, Βρυξέλλες. Υπάρχει το πρόγραμμα της γεωγραφικής κατανομής. Σουηδία, Δανία, Γερμανία. Αυτοί δεν θέλουν να έρθουν, ε. γιατί ξέρετε κάτι, αν είσαστε διευθυντής Υπουργείου στο Μόναχο και ο ε, ή αν θέλετε διευθυντή σε, μία τράπεζα και έχετε δύο παιδιά, το να έρθετε στις Βρυξέλλες στο Λουξεμβούργο δεν αξίζει, δεν έρχονται. Και ξέρετε κάτι, τώρα είμαστε και αναγκασμένοι να κάνουμε και εκστρατεία προσέλκυσης ανθρώπων, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε, θα γίνει στη Βουλγαρία, στην ε, Κομισιόν, στην, ε, στις Βρυξέλλες, θα έχουμε ε, τους Βούλγαρους που θα θέλουν μόνο αυτοί να έρθουν στις Βρυξέλλες αλλά είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην εκπλαγούμε στο τέλος ότι θα υπάρχουν κράτη που δεν θα θέλει κανείς, μα κανείς να έρθει στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, υπάρχουν και δύο βασικά θέματα. Το νυν δημοσιονομικό πλαίσιο εγκρίθηκε πολύ κατηστερημένα. Το Δεκέμβριο του 2013 ε, είχε καταστεί σαφές ότι τότε θα έπρεπε να υπάρχουν τα partnership agreements. Δηλαδή η Κομισιόν διαπραγματεύεται με υπουργού περιβάλλοντος, ε, κοινωνικών υποθέσεων, ε, υποδομών, οικονομικών. Και αυτό διαρκεί ένα χρόνο. Αυτές οι συμφωνίες ε, πρέπει να εγκριθούν καταρχήν σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου λόγω της συγχραματοδότησης. Έτσι λοιπόν έχουμε προγράμματα που αρχίζουν να τρέχουν που άρχισαν να τρέχουν, γιατί ξεκίνησαν το 2013 όπως σας είπα, το 2015 άρχισαν να τρέχουν τα πρώτα προγράμματα. Και αν ισχύει ο τύπος N συν 3, ε, τότε θα είναι δυνατόν η η λογαριασμοί να υποβληθούν πολύ καθυστερημένα, πολύ αργότερα από τη στιγμή που γίνεται η επένδυση. Και γι' αυτό εμείς λέμε όχι, να πάμε πίσω στο 1 συν 2 και ελπίζουμε ο προπολογισμό να έχει εγκριθεί μέχρι το τέλο του έτου, έτσι ώστε την πρώτη η του επόμενου έτου, με έγκριση κονδυλίων, να μπορούμε να περάσουμε στην εκτέλεση του προπολογισμού. Σε λίγες μέρες ε, θα δώσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών την έκθεση για τα ραλ. Αυτό το κάνουμε τρεις φορές το χρόνο και θα το κάνουμε τώρα εντός λίγων εβδομάδων. Όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματο. και για αυτά είμαστε σε επαφή με το ελεγκτικό συνέδριο για να καταλήξουμε σε ένα κοινό ορισμό. Γιατί χρειαζόμαστε και προσωρινό και τελικό ε, ορισμό ο προσωρινός λέει πού κάναμε λάθος, πού, πού μπερδευτήκαμε στους ε, λογαριασμούς, κάναμε λάθος ενδεχομένως στους ελέγχους ή πού ε, εντοπίσαμε απάτες, ε, καταχρήσεις, απιστίες. Αυτά είναι οι πρώτοι υπολογισμοί λάθους που μπορεί να έχουν λάθη στην Κομισιόν ή στα κρατημέλη ή και στους δύο. Όμως για τον φορολογούμενο είναι πολύ σημαντικότερο το τελικό ποσοστό λάθος σφάλματος. Γιατί αυτό που εντοπίζουμε με αυτό, από αυτό ωφελείται ο ε, πολίτης. Πρέπει λοιπόν να ισχύουν και οι δύο ορισμοί να εξετάζετε εσείς ε, την ποιότητα της δουλειάς μας και ο φορολογούμενος να γνωρίζει ποια είναι τα χρήματα τα οποία έχει χάσει. Γιατί ε, καταθέτουμε διορθωτικό προϋπολογισμό. Ε, ποια ε, κονδύλια χρειάζονται. Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία λένε ότι ας πούμε το 2019 χρειάζονται νυν χι κονδύλια και ε, τα κονδύλια που ζητήθηκαν αυτά θα πρέπει να αντιστοιχούν με τα απαραίτητα κονδύλια. Κατά το παρελθόν πολλά κράτη ζήταγαν περισσότερα κονδύλια και επειδή καθυστερούσαν στους διαγωνισμούς ε, ε, στην ανάθεση έργων, ε, τα κονδύλια που είχαν αισθηθεί ήταν περιτά, δεν χρειαζόντουσαν. Φέτος όμως με το διορθωτικό μας προπολισμό δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους θέμα. Τι θα γίνει αν έχουμε Brexit χωρίς συμφωνία. Κάθε μέρα το ζούμε αυτό. Ε, πραγματικά μας εντυπωσιάζει ο κύριος Τζόνσον κάθε μέρα με τις δηλώσεις του και χαιρόμαστε που τελικά το Κοινοβούλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο κάπως αρχίζουν να συμπλέουν. Αν τελικά υπάρξει αποχώρηση τέλειο Οκτωβρίου χωρίς καμία απολύτως συμφωνία και η κυβέρνηση ε, κάνει αυτό που έχει πει ότι δεν θα επιστρέψει και δεν θα πληρώσει τίποτα, θα πρέπει από την 1η Νοεμβρίου να κλείσουν. Να διώξουμε τα παιδιά που είναι στο Εράσμους να πάνε πίσω ε, στην ε, Βρετανία. Δεν θα χρηματοδοτεί ούτε η Οξφόρδη ούτε το Κέμπριτζ. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μεταξύ κάποια λύση θα βρεθεί για τον προπολογισμό. Το 2019 έχει κλείσει, θα μας ε, λείψει περίπου ένα δις, ε, κάπως θα το καλύψουμε αυτό. Όμως σας έχει κατατεθεί το σχέδιο του προπλογισμού, έχει ξεκινήσει ε, ο τριμερής διάλογος, ε, η συνδιαλλαγή θα ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου. Αν φύγουν οι Βρετανοί μετά από τρεις μέρες, στις 31, αυτό θα, είναι, ε, θα σημαίνει ότι θα μας λείπουν 12 δις. Και επειδή το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το μόνο που δεν μπορεί να κάνει χρέη, σε αντίθεση με τα κράτη-μέλη και την τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να κλείσουμε το κενό αυτό εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εγώ λέω, βεβαίως εσείς τα αποφασίσατε, Είμαι σε επαφή με την Επιτροπή Προϋπολογισμών για το δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης δεκαετίας, εγώ προτείνω το εξή για την έλλειψη του Brexit. Το μισό να ε, το καλύψουμε με περικοπές και το άλλο μισό με μεγαλύτερες εισφορές. Για το επόμενο, την επόμενη δεκαετία. Νομίζω αυτή είναι η λύση και γι' αυτό περίπου κατά τις 15-18 Οκτωβρίου θα πάω στο Κολέγιο των Επιτρόπων, το αργότερο μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να καταθέσω, να προτείνω διορθωτικό προπολογισμό που θα πρέπει να σας έχω δώσει πριν από τις συνδιαλλαγές και εκεί θα λέω 5,5 δις ε, πληρωμές και 5,5 δις ε, περικοπές. Ε, αλλά δεν ξέρω νομικά δεν μπορούμε να κόψουμε τις πληρωμές ε, για τους γεωργούς, γιατί αυτά που θα πάρουν του χρόνου θα εξαρτώνται από το φετινό αποτέλεσμα. Εγώ λοιπόν ε, δεν θέλω να προκαλέσω ζημιές ε, και γι' αυτό το λόγο θα επανέλθω κατά τα μέσα τέλη Οκτωβρίου σε εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το θέμα του προσωπικού, ε, έχουμε όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα Λουξεμβούργου. Υπάρχει η συνθήκη, λέει ε, πόσοι θα πρέπει να εργάζονται στο Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο το κόστος ζωής είναι υψηλό, 10% ε, 100 ψηλότερα ενίκεια. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε το Λουξεμβούργο να παραμείνει ένας χώρος ελκυστικός για νέους ε, και κυρίως για αυτούς που έχουν οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αλλά επίσης ε, και για την επιβεβαίωση της αγαστής μας συνεργασίας. Αλλά να σας πω κάτι, δεν με ξεφορτωθήκατε, άλλες δύο φορές θα έρθω εδώ. Στις 18 Δεκάτου θα έρθω στο Στρασβούργο, στην και αν δεν δεχτείτε τον υποψήφιο, τον πρωτό υποψήφιο, θα με λουστείτε μέχρι τα Χριστούγεννα. Ε, υπάρχει και το θέμα των, του Αντιπροέδρου για το EMG. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Το πρώτο ε, έχει ήδη ληφθεί υπόψη, θα το σεβαστούμε. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα κάποιες πληροφορίες και κάποιους αριθμούς ε, από το ΙΝΚΕ. Ε, μόλις πάρουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία, τότε θα εφαρμόσουμε την απόφαση και θα είμαστε ε, αξιότιμος εταίρος. Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πληρέστατη η επισκόπηση και απαντήσεις σας πληρέστατες. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό σφάλματος, όμως, αν έχουμε δύο από το ελεγκτικό και δύο από εδώ, ε, κάτι δεν πάει καλά. Πού είναι το πρόβλημα, πού υπάρχουν οι δυσκολίες. Μπορεί να μην είναι μόνο στην Κομισιόν, μπορεί να είναι στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας αν υπάρχουν δυνατότητες ε, απάτης και αν υπάρχουν πρέπει να κλείσουμε τις τρύπε και τα κενά, τα παραθυράκια. Και αυτό πραγματικά το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι ε, βλέπουμε να ανακύπτουν συνεχώς νέες απαιτήσει ε, και νομίζω ότι θα πρέπει και το ελεγκτικό και η Κομισιόν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Σε ό,τι αφορά την περισσότερικού ελέγχου, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι και ο ε, Γενικός Διευθυντής, στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση, Γενικό Διευθυντή ε, τη ε, υπηρεσία μα μίλησε για 13 διαφορετικά ποσοστά σφάλματο. Ε, δεν είναι λίγο πολύπλοκο, δεν ξέρω, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι πιο λογικό κάποιες λιγότερες ε, τέτοιες, λιγότερα ποσοστά να δίνονται. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος άλλος έχει να είσαι ερώτηση στον Επίτροπο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Άρα, να αποχαιρετήσουμε τον Επίτροπο που έχει πολλά να κάνει και να κρατήσουμε λίγο μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή. Ähm, wir haben ja, äh, Generaldirektor,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 Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε ο Επίτροπο Σέτιγκερ, κατ' η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγή την έκθεση για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο και τις συστάσεις που ε, ακολουθούν. Αυτή η δημόσια έκθεση αποδεικνύει, θα έλεγα, την αφοσίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον έλεγχο και στην διαφάνεια προσπαθούμε να δείξουμε με απόλυτα διαφανή τρόπο τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε και τις αδυναμίες τους επίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αναλαμβάνει και πολύ ε, σημαντικές δράσεις για να κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις. Δίνουμε ε, συστάσεις και ενημερωτικά στοιχεία στο πρώτο τμήμα του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βλέπετε ότι υπάρχει ένα έγγραφο που έχει ενσωματωθεί, το οποίο περιγράφει ακριβώς τις πρόσφατες δράσεις του 18. Πριν σας δώσω περισσότερες πληροφορίες τώρα για τα αποτελέσματα ε, και, την, ε, και το εύρος του λογιστικού ελέγχου, θα ήθελα να σας πω ακριβώς ποιο ήταν το πλαίσιο του λογιστικού ελέγχου το 18. Από την 1η Ιανουαρίου του 18 το 100% των πιστώσεων είχαν απορροφηθεί. Στο σύνολο το IS περιελάμβανε 166 δράσεις, 48 λογιστικοί έλεγχοι, 140 εκ των υστέρων έλεγχοι, δύο περιορισμένες αναθεωρήσεις και δύο διαβουλευτικές συναντήσεις. Ήδη από το 2015 έχουμε δημοσιεύσει 233 συστάσεις. Όπως είπε ο κύριος Σέτιγκερ, το 100% έγιναν αποδεκτές. Όλες οι αναθεωρήσεις αυτές ήταν επί τη βάση ε, προσχεδίων τα οποία είχαν γίνει δεκτά ανατομέα από τον EIS. Απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή των συστάσεων αυτών, ω εκ τούτου δεν έχει νόημα να μιλήσω για την εφαρμογή τώρα των συστάσεων, οι οποίε έγιναν αποδεκτές το 2018. Δεν υπάρχει αρκετός ενδιάμεσος χρόνος, γι' αυτό θα ήθελα να σας δώσω το τι συμβαίνει με το λεγόμενο follow-up. 1938 συστάσεις μέχρι το 15. 572 εφαρμόστηκαν, το 81% λέει ο Επίτροπος. Υπάρχει μία εφαρμογή κατά 90% και το 5,3% γύρω στις 100 αγνοήθηκαν ουσιαστικά. Μόνο το 2,9 όμως τελικά των κρίσιμων και ιδιαίτερα σημαντικών συστάσεων δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Υπάρχει μια καθυστέρηση δηλαδή άνω των 6 μηνών σχετικά με την αρχική προθεσμία εφαρμογής. Το δεύτερο τμήμα τώρα του εγγράφου εργασίας ε, για το προσωπικό της Επιτροπής δίνει α, συγκεκριμένα στοιχεία για το λεγόμενο follow-up. Το EIS θεωρεί ότι τα στάδια εφαρμογής των συστάσεων των λογιστικών ελέγχων είναι συγκρίσιμο με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει προσοχή σε 18 πολύ σημαντικές καθυστερημένες συστάσεις ε, και λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο τρίτο τμήμα του εγγράφου εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής. Να περάσω τώρα στα συμπεράσματα επί τη βάση των λογιστικών ελέγχων του 2018 και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω την προσοχή σας σε δύο πλευρές της εσωτερικής λογιστικής προσπάθειας. Πρώτον, το EIS σε σχέση με τις επιδόσεις και δεύτερον η σύσταση για την χρηματοπιστωτική, χρηματοοικονομική συγγνώμη, διαχείριση για τις επιδόσεις. Ε, σύμφωνα και με τον, με τον οικονομικό κανονισμό και την χάρτα του EIS, Ζητήσαμε από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές να μας βρουν τους χώρους βελτίωσης. Οι εσωτερικοί έλεγχοι συγκέντρισαν την προσπάθειά τους το 2018 σε τομείς όπως οι συνέργειες, βελτίωση αποτελεσματικότητα, διακυβέρνηση, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και προσμέτρηση επιδόσεων στα πλαίσια της εφαρμογής του προϋπολογισμού στις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άμεσες, έμεσες και ε, μοιρασμένης ε, κατανομής. Υπήρξαν σημεία στα οποία θα πρέπει να υπάρχει βελτίωση και επίσης είδαμε ότι υπάρχει βελτίωση ήδη σε κάποιους άλλους τομείς. Τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται. Τα συγκεκριμένα αυτά προγράμματα δράσης ανταποκρίνονται στα αιτήματα των λογιστικών μας ελέγχων όπως αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί από το EIS. Το πρώτο τμήμα του εγγράφου περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις συγκεκριμένες αποστολές. Έρχομαι τώρα στην γνωμοδότηση EIS για την χρηματοοικονομική διαχείριση. Ως προς την πλευρά αυτή θα ήθελα να σας υποχραμίσω ότι εμείς έχουμε εκδώσει μια γνωμοδότηση για το σύνολο των επιδόσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής που βασίζεται σε συνολικούς λογιστικούς ελέγχους τους οποίους έχει αναλάβει η ΑΕΣ όπως επίσης και σε εκθέσεις ε, που προέρχονται από το ελεγκτικό συνέδριο για το λογιστικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι συναλλικά τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου της Επιτροπής είναι λειτουργικά. Υπάρχουν τομείς όμως όπου ορισμένες αδυναμίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Ως εκ τούτου λοιπόν εκθέτω για μία ακόμη φορά τη θετική μου γνώμη η οποία είναι τεκμηριωμένη και από τις επιφυλάξεις οι οποίες είχαν γίνει για την έκθεση την αναλυτική και τις δηλώσεις των Γενικών Διευθυντών του 18 έλαβα υπόψη τα συνδυασμένα αποτελέσματα των συνολικών ποσών που χρησιμοποιήθηκαν ε, και τις διορθώσεις που έγιναν από τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου, κάτι το οποίο δείχνει ότι ο νέος προϋπολογισμός είναι κατάλληλα προστατευμένος και ποσοτικά και χρονικά. Και αναφέρθηκε σε αυτό ο Έτιγκερ. Δεν λέω ότι τα πάντα είναι τέλεια. Εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες και βελτιώσεις ακόμα πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά το σύστημά μας είναι λειτουργικό και αποδίδει. Έχουμε όμως ενταπίσει τα προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο όμως πρέπει να υπογραμμίσω και το οποίο έχω εντοπίσει και υπογραμμίσει και τα προηγούμενα χρόνια, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερα έμφαση. Σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών ταμείων, αναφέρομαι στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαρτάται από την εφαρμογή ενδιαμέσων άλλων σωμάτων τρίτων χωρών, σαν παράδειγμα διεθνών οργανισμών, εθνικών υπηρεσιών, κοινών υπηρεσιών, σωμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συγκεντρωτικών οργανισμών. Για να μπορέσουν όλοι να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ελέγξει την εφαρμογή των προγραμμάτων και από πλευρά των εταίρων αυτών. Οι γενικές είναι πόσο πρέπει να ορίσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες μορφές παρακολούθησης των παράπλευρων αυτών δραστηριοτήτων έτσι ώστε οι λειτουργούσες κατ' εξουσιοδότηση αυτές οι υπηρεσίες να προστατεύουν και αυτές με αποτελεσματικό τρόπο τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το feedback το οποίο έχω πάρει από τους λογιστικούς ελέγχους που έκαναν οι υπηρεσίες μου για τους διαφορετικούς αυτούς εταίρους δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εταίρων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό να υπογραμμίσω ότι τα συμπεράσματα των λογιστικών μας ελέγχων ασχολήθηκαν και με, ε, σε υψηλό επίπεδο υπαλληλικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει η Επιτροπή ε, ε, Λογιστικού Ελέγχου που αποτελείται από έξι επιτρόπους και τρία εξωτερικά μέλη. Η Επιτροπή αυτή εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο και δίνει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των συστάσεων των προηγούμενων λογιστικών ελέγχων από τις Γενικές Διευθύνσεις. Κλείνοντας να πω ότι και η Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου και η Επιτροπή Βελτίωσης του Λογιστικού Ελέγχου έφεραν εις πέρα στην αποστολή τους έτσι ώστε τα συστήματά μας να λειτουργήσουν σωστά και εντόπισαν τις αδυναμίες έγκαιρα και με ακρίβεια. Υπάρχουν θετικά στοιχεία σε πάρα πολλούς τομείς. Θα έλεγα ότι σε όλους τους τομείς στους οποίους είχαν παλιότερα αντιμετωπιστεί αδυναμίες. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει βελτιωθεί τα προηγούμενα χρόνια και είμαι πεπισμένος ότι επί τη βάση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του 18, όπως επίσης και στην παρακολούθηση όλων των συστάσεων και των προγραμμάτων δράσης από τα EPC, τα συστήματά μας συνολικά βελτιώθηκαν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά για την διεξοδικότατη παρουσίαση. Ξεκινήσω εγώ με τις ερωτήσεις καθότι είμαι συγγήτρια. Υπάρχουν τα λεγόμενα ευρεδικά έργα της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΙΕΡ. Hybrid projects. Εγώ δεν είμαι πολύ έμπειρη ε, και ρώτησα πιο μέσα από που και αυτοί ξέρουν το κεφάλι τους. Δεν μπορείτε να μα εξηγήσετε τι είναι αυτό το υβριδικό project. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα περί τίνο πρόκειται. Κανένα δεν με διεφώτισε επ' αυτού. Δεύτερο, Μια ερώτηση που θέλω να ρωτήσω, να κάνω. σε ό,τι αφορά τις πηγές φαλμάτων ή ε, ενδεχόμενης απάτης ή άλλων αξιόπινων πράξεων ε, εσείς από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πού εντοπίζετε ε, αυτές τις πηγές κυρίως. Υπάρχει σίγουρα και μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος που έχει ως αποτέλεσμα οι υποβάλλοντες αίτηση να μην ξέρουν ποιο είναι το επιλέξιμο κόστος. Είναι πολύ πολύπλοκες οι λίστες με τα κριτήρια, πρέπει να κάνουν προβολές ε, και, και άλλες ε, μελέτες και υπολογισμούς πριν καταλήξουν ε, στις αιτήσει τους. Ο βαθμός λοιπόν αυτή τη γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας επηρεάζει και αν ναι πόσο τα σφάλματα και επίσης αν υπάρχει δυνατότητα να περιορίσουμε, να αποτρέψουμε κλιματικές δραστηριότητες μέχρι σε προσωπικό χρηματισμό, σύγκρουση συμφερόντων ε, ή ε, άλλες ε, παράνομες ενέργειες. Επίσης, το είπα και στον Επίτροπο, έτσι προσεκτικά του το ερώτημα, γάμα δέλτα μάρε ρέγγιο. 13 διαφορετικά ποσοστά σφάλματος πρέπει να τα βγάλουν πέρα και αυτό είναι πολύ πολύπλοκο. Γιατί μετά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι σφάλμα, τι δεν είναι σφάλμα, ούτε πού εντοπίζονται τα προβλήματα. Και αυτό δυσκολεύει το έργο μας. Τελευταία ερώτηση για το follow-up των εκκρεμουσών υποθέσεων στην όλα. Αυτή κάνουν υπηρεσίες σας για την επανόρθωση και την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων σε διάφορες ε, γενικές ε, διευθύνσεις όπως είναι η RD, DEFCO, Apple και τα λοιπά που μιλάνε για κάποιο πρόβλημα στην ευαισθητοποίηση και για την πρακτική εφαρμογή του EDS. Ich gehe vielleicht die. Äh, Δεν υπάρχουν ερωτήσεις από την ε, ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Άρα ο Ολιβιέ θα πάρει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ε, συγχαρώ ε, την Υπηρεσία Ιστορικού Ελέγχου τη Κομισιόν για το κολοσιαίο έργο. Το βλέπουμε ε, από την έκθεση με τον αριθμό των προγραμματισμένων και πραγματοποιηθέντων ελέγχων, παρακολούθηση των δράσεων, των διορθωτικών που προτείνεται κτλ. Πολύ σημαντική δουλειά που επιτρέπει τη διόρθωση ορισμένων καταστάσεων ε, πολύ πριν ε, ε, περάσουν στην εκτός κομισιών και γίνουν ευρύτερα τα προβλήματα και μεγαλύτερα. Δύο ερωτήσεις. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει γενικότερα με το μηχανισμό, το θεσμικό, τον επιχειρησιακό της διακυβέρνησης που έχει κάποιες αδυναμίες ακόμα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση ως διευθυντή αυτής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν θέλησε και τελικά κατάφερε ή δεν κατάφερε να βελτιώσει του μηχανισμού διακυβέρνηση. Δεύτερο ερώτημα, Όλαφ. στο πλαίσιο αυτού του συστήματο προφορική έχουμε διάφορε λεπτέ ε, πληροφορίε, ευαίσθητε. Η Όλαφ μα λέτε ότι εφαρμόζει καλέ πρακτικέ για να μειώσει του κινδύνου ασφαλεία ε, σε ό,τι αφορά την πληροφορική, επαναλαμβάνω. Γνωρίζουμε ότι το σύστημα διαχείριση των περιεχομένων είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί. Ένα ακρογωνιαίο λήθο για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά τη η υπηρεσία. Τι ε, έχετε να μα πείτε. Αυτή η πληροφορική ασφάλεια, πώς λαμβάνετε υπόψη από την Όλαφ. Έχετε μήπως ε, κάποιες συμπροματικές συστάσεις πέραν των όσων ε, ήδη έχουν εφαρμόσει. Εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Ή ναι. Ναι, ο Πέτρη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ψιλοδίσταζα, γιατί δεν και τόσο εντός θέματος, αλλά αφού έχω τη δυνατότητα στον ε, αξιότιμο Γενικό Διευθυντή, ε, τον κύριο Καφ, να μην τη χάσω και να του κάνω την ερώτηση που θέλω σε ό,τι αφορά τα χρήματα που περνάνε από τα χέρια σας, ε, από την Κομισιόν και βλέπουμε χρηστή διαχείριση σχεδόν στο 100%. Αλλά τι έχετε να μας πείτε. Say, you know, to anyone... Όποιος κοιτάζει εκτός, ε, από, από έξω, τι κάνουμε εμείς εδώ, πρέπει να εκπλήσετε προσπαθώντας να καταλάβει ε, και να προβληματίζεται, προσπαθώντας να καταλάβει πώς μπορεί η Κομισιόν τέλος πάντων να ελέγξει και να παρακολουθήσει την τήρηση όλων των κανόνων κατά τη χρησιμοποίηση των ε, κονδυλίων. Αφού η Κομισιόν βασίζεται, πρέπει να βασιστεί, δεν έχει άλλη επιλογή, στα στοιχεία που στέλνουν τα κράτη-μέλη και είναι κάπως αμφισβητούμενη η διαφάνεια. Εσείς μπορείτε να μας πείτε ναι. Έτσι έγιναν τα πράγματα, αλλά οι φορολογούμενοι ε, θεμητά ανησυχούν και δίκαια ανησυχούν. Γιατί δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι είναι 100% αξιόπιστα τα στοιχεία που σας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχει μια ομίχλη γύρω από όλο τον τρόπο με τον οποίο δαπανά το προπολογισμό. Ευχαριστώ. So my to you... Άρα, τώρα έρχομαι στο ερώτημά μου σήμερα. Νομίζω ότι πολλές φορές σας το έχουν ξαναθέσει, αλλά θα σας το ξαναθέσω σήμερα εγώ. Τι πρέπει να γίνει με αυτό. Nun darf ich Herrn Generaldirektor um seine Antwort bitten. Να παρακαλέσω τον Γενικό Διευθυντή να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ξεκινήσουμε με τις δικές σας ερωτήσεις. Δυστυχώς ε, πρέπει να σας πω ότι την ε, πρώτη σας ε, ερώτηση δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Αυτά τα γάμα δέλτα near hybrid projects ούτε και εγώ τα ξέρω. Ε, ούτε και εγώ έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Πάντω θα ενημερωθώ και γραπτό θα σα απαντήσω για τα, τα αυτά που πρέπει. Ε, λοιπόν, με ακούλπα. Αυτό με καθισκάζει λέει η κυρία Χολμάρη, που δεν ξέρετε κι εσεί. Ναι, είστε, έχετε καλή παρέα εδώ. Δεν είστε οι μόνοι που δεν καταλαβαίνετε τι θα πει υβριδικό σχέδιο. Λοιπόν, πάω στο επόμενο ερώτημα που είναι σημαντικό. Εν ολίγης, ουσιαστικά με ρωτάτε οι υψηλότεροι κίνδυνοι που εντοπίζονται και τι μπορούμε να κάνουμε για να τους διαχειριστούμε. Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά σφάλματο. Εδώ θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα με το ελεγκτικό που λέει όπως και εμείς ότι εδώ και κάποια χρόνια η πηγή σφαλμάτων είναι, όπως είπατε και εσείς, οι πολύπλοκοι κανόνες και μας δεν ξεκάθαρα. Όταν Κομισιόν και εταίροι συνεργαζόμαστε για τους κανόνες επιλεξμάτων που είναι πολύπλοκοι, Εκεί βλέπουμε και ε, πολύ ψηλά ποσοστά σφάλματος. Επίσης, οι πληρωμές βασίζονται σε σημαντικές προϋποθέσεις και όρους. Στην πραγματικότητα όμως αυτό οδηγεί στο εξής. Ναι, με να έχουμε κάτω του δύο... Ε, ποσοστό σφάλματος για το συγκεκριμένο αυτό προπολογισμό, ενώ στο άλλο τμήμα του προπολογισμού να έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά σφάλματο. Άρα απλούστευση. Αυτό είναι το κλειδί για μένα. Θέλουμε περισσότερη πρόοδο. Και νομίζω ότι μα δίνεται τώρα μια πολύ καλή δυνατότητα και ευκαιρία. Για ποιο λόγο, διότι το νέο πλαίσιο, διότι το νομικό πλαίσιο για το πολιετέ δημοσιονομικό, για την πολιετή φάση εφαρμογής ε, του προπολογισμού θα ολοκληρωθεί του επόμενου μήνες από εσά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαιτέρως. Απευθύνω έκκληση και εκ μέρου όλων των συναδέλφων στην Κομισιόν. Παρακαλώ, βοηθήστε μας να προχωρήσουμε σε όσο το μεγαλύτερη απλούστευση των κανόνων, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν πιο εύκολα να συμμορφούνται προς τους όρους και τους κανόνες. Και έτσι όλοι στο σύστημα θα μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει. Νομίζω ότι έχουν ήδη γίνει πολλά από την Όλαφ σε συνεργασία με τους εταίρους. Όπως ξέρετε υπάρχει αυτή η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης. Ε, ήταν εδώ ο Γενικός Διευθυντής Όλαφ, ε, εξήγησε τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και το τι απομένει να γίνει. Νομίζω ότι σε καλό δρόμο βρίσκεστε και σε ό,τι αφορά τον αριθμό ε, εικαζόμενων απατών που και μάλλον που έχουν εντοπίσει εξωτερικά και εμείς είναι πολύ περιορισμένος. Φυσικά και μία τέτοια περίπτωση να πληρωθεί είναι κακό. Αλλά δεν παραγνωρίζουμε τον κίνδυνο, προσπαθούμε να τον αντιμετωπίσουμε, να τον διαχειριστούμε, ώστε να μείνει σε αποδεκτά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά τους πολύ διαφορετικούς ε, τύπους ε, και ορολογίες που χρησιμοποιούνται από γάμα δέλτα ρέγγιο μάρ και, ε, και άλλες μπορείτε να προσθέσετε γενικές διευθύνσεις. Ποια είναι η λύση, ποια είναι η εξήγηση. Θέλουν ουσιαστικά στους ενδιαφερομένους να δώσουν τις καλύτερες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στα συστήματα. Βέβαια θα μου πείτε και το πολλό το F σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί να μην συγκεντρωθούμε στα βασικά για να διευκολύνουμε το έργο μας, την κατανόησή μας, ε, το έργο και των ε, ελεγκτών. Εμείς στην εσωτερική υπηρεσία εστιάζουμε σε δύο σημεία. Τα είπε ο Επίτροπος Έτιγκερ. Το πρώτο είναι ε, το κίνδυνος για τις πληρωμές, ποσοστό φάλματος, Άπαξ και δώσουμε εντολή, έγκριση για να γίνει μια πληρωμή. Ποιο είναι το πρόβλημα και στο κλείσιμο ποιο είναι, ποιος είναι ο κίνδυνος. αφού ολοκληρωθεί το έργο μας και έχουμε κάνει τις οικονομικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις, ποιο είναι το ποσό που παραμένει παράνομο εντό αγωγικών. Βέβαια, εδώ έχουμε και τις εκτιμήσεις. Στηριζόμαστε σε πολλούς τομείς στα δεδομένα που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Τα βασικά δεδομένα των κρατών μελών, παραδείγματος χάρη στα διαφθορτικά ταμεία ή στη γεωργία, είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία που σας δίνει το ελεγκτικό συνέδριο βάσει στατιστικού δείγματος και προεκβολής. σε σχέση με όλο τον πληθυσμό. Για τον κύριο Σαρβαμά. Τι κάνουμε όταν δεν μας δίνουν αξιόπιστα στοιχεία τα κράτη-μέλη. Ή γιατί η δειγματοληψία δεν ήταν σωστή, ή δεν κάνανε σωστή παρεκβολή, παρεκβολή δεν βρήκαν όλα τα σφάλματα. Εμείς τι κάνουμε τότε. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα ρεαλιστικό ποσοστό σφάλματος. Δηλαδή το στατιστικό δίκτυ τον αντικαστούμε την προσωπική μας κρίση ουσιαστικά και παίρνουμε υπόψη όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και καταλήγουμε σε ένα κατεκτήμηση ποσό. Χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση να είναι μια μηχανική προσέγγιση. Εδώ συμμετέχει προσωπική κρίση, επαγγελματική κρίση. Τώρα, συνεργασία και το ίντες. Έχουμε εντοπίσει προβλήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη γνώση ε, εκ μέρους των συναδέλφων. Δηλαδή, ποιοι είναι οι κανόνες και πώς εφαρμόζονται. Οπότε και συνιστούμε περαιτέρω επιμόρφωση με εκπαίδευση. και θα βελτιωθεί αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τα κοπλιμέντα για το κολοσσίο έργο που είπατε της ε, Γενικής μου ε, έχετε δίκιο ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Είναι πολύ κολοσιαίο και πολύ σημαντικό το έργο που κάνουμε. Κάνατε μια ερώτηση συγκεκριμένη για τη διακυβέρνηση. Πρέπει να σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά την έκθεση που ήταν ε, ουσιαστικά συνέχεια μια ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ε, προδιετία τριετία. Εμεί κάναμε έναν έλεγχο ε, λογιστικό και διατυπώσαμε συστάσεις για τη βελτίωση τη διακυβέρνηση. Παραδείγματο χάρη σε επίπεδο τη επιτροπή Προόδου του ΕΛΕ ή στο επίπεδο ανάλυση κινδύνου και πολλά άλλα στοιχεία αναφέραμε. Μπορώ να σα πω λοιπόν κύριε Βουλευτά Πώ όλε οι συστάσει μα υλοποιήθηκαν Υπήρξε σχέδιο δράσης συγκεκριμένου. Πριν από κάποιες εβδομάδες ε, το κλείσαμε, που σημαίνει ότι είχαμε, ε, καταφέραμε να επηρεάσουμε. Και το ίδιο μπορώ να πω για τη διακυβέρνηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Εδώ η πρόταση είναι τεράστια. Βέβαια, μένουν ακόμα να γίνουν κάποια πράγματα, είμαστε όμως στο σωστό δρόμο. Που σημαίνει ότι τα πορίσματά μας λαμβάνονται υπόψη. σε σχέση με το ερώτημα του κυρίου Σαρβαμά για το πώς ελέγχεται ε, όλο αυτό το χρήμα που περνάει τα συστήματά μας, δηλαδή ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες και ότι είναι όλοι και όλα αποδοτικά αποτελεσματικά. Αυτό σχετίζεται με την ε, αιμονή που έχω ε, να υπάρχει σωστή εφαρμογή της μεθόδου, άλλο βέβαια η μεικτή διαχείριση και άλλο η δική μας διαχείριση. Αλλά πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να υπάρχει ε, ε, σωστός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου. Όποτε δηλαδή προκύψει κάποιο πρόβλημα, εμείς λαμβάνουμε, αναλαμβάνουμε δράση αλλά αν εξακολουθούν να μην λειτουργούν τα συστήματα και να παρουσιάζουν αδυναμίες, τότε πρέπει να επιβάλλουμε χρηματοοικονομικές διορθώσεις. Μπορώ να σας ε, ενημερώσω με τα χαράς ε, για το ότι επειδή θα παρουσιάσω την επόμενη εβδομάδα στο Ζάγκρεμπ ε, όπου θα έχω του ομολόγους από την συνοχή για να συζητήσουμε το πώς εφαρμόζεται ο προπολισμός της Ένωσης στον τομέα της συνοχής, για να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει θα μιλήσω ηλική λοιπόν και θα πω τι μπορούμε να κάνουμε για τη βελτίωση. Όσο κάθεται ο Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, δράτω με τη ευκαιρία. Ακούστε. Το ερώτημά μου αφορούσε κάτι που εγώ, εσεί, εμεί δεν γνωρίζουμε καν. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αν δεν ξέρουμε αν το χύψη κράτο μέλο. σκοπίμως ή όχι δεν δίνει αξιόπιστα στοιχεία. Τα βάζει σε άλλη κατηγορία, από εκεί που θα έπρεπε, για παράδειγμα, κάποια στοιχεία. Από τη στιγμή αυτή και μετά υπάρχει λάθος ενημέρωση. Και εσεί όταν φτάσουν τα στοιχεία στα χέρια σας, ούτε καν ιδέα έχετε ότι δεν είναι σωστά αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα το οποίο εννοώ και που αυτό με προβληματίζει κάθε χρόνο. Δεν ξέρω, ίσως να μην τα απάντηση σήμερα γιατί αν είχατε δεν θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, ε, να προσθέσω κάτι κύριε Κράφτε. τίτε το ερώτημα και πολλοί λένε ότι γυρίζουμε γύρω από τον ίδιο μας τον ίσκιο, ότι ε, κάποια στιγμή τα ποσοστά σφάλματος ε, δεν αλλάζουν όπως θα το θέλαμε, αλλά σε τελική ανάλυση ε, δίδονται χρήματα όχι για το στόχο που έχουμε θέσει, αλλά τα χρήματα τα παίρνουν τα κράτη-μέλη ε, τα παίρνουν λοιπόν για τον εαυτό τους. Για μένα λοιπόν τίθε το ερώτημα. Σε ένα μελλοντικό ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε τα εθνικά χαρτοφυλάκια, τα envelopes και εάν διαπιστώσουμε ότι το ποσοστό ασφάλματος ξεπερνάει το 3 ή 4%. Μήπως θα είχε νόημα τότε στην περίπτωση αυτή με ειδικό προσωπικό το οποίο θα το στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθούμε γιατί τότε θα υπήρχαν περισσότερες δυνατότητες ε, οι ε, ετούντες να μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο τους. Δεν θα ήταν καλύτερα αυτό από το να διαμετρώμεθα μετά από πέντε χρόνια. Ε, το ρωτάω απλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση και τον κύριο Ζαμαβά επίσης για την ερώτηση. Θέλω να σας πω ότι τα συστήματα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζονται στο να ελέγξουμε το κατά πόσον τα κράτη-μέλη που μας δίνουν τα στοιχεία είναι σωστά ή όχι. Αν δεν είναι σωστά πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και ε, με ε, τα πολιτή πλαίσια ε, δεν το καταφέρνουμε αυτό απόλυτα. Γι' αυτό λοιπόν γνωρίζω ότι είσαστε υποπίεση χρόνου. Πολύ σύντομα λοιπόν κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας πω, δέστε λιγάκι την έκθεση της ετήσια διαχείρισης και οικονομικών επιδόσεων. Εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο που αφορά τον, την προστασία του ενωσιακού προεπλογισμού και εκεί βλέπετε ακριβώς ε, πώς γίνονται οι διορθώσεις σε κάθε κράτος μέλος ε, στα πλαίσια της διαχείρισης κονδυλίων και δέστε λιγάκι ε, τι γίνεται με τα απόλυτα ποσά. Ε, έτσι θα έχετε κάποιους δείκτες που τα αφορούν στον κίνδυνο. Και εσείς ε, στην περίπτωση αυτή ως πολιτικός έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε μέτρα και να παρακαλέσετε μας να ελέγξουμε το κατά πόσον με τα μέτρα που προτείνετε μπορούν να επιτευχθούν διορθώσεις. Νομίζω όμως ότι ο Επίτροπος ανέφερε τον αριθμό των προγραμμάτων και είναι μη ρεαλιστικό το να πιστεύει κανείς ότι οι ενωσιακοί υπάλληλοι μπορούν να αντικαταστήσουν τους εθνικούς υπαλλήλους για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων. No other alternative than really to have a sound monitor. Δεν υπάρχει άλλη. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια σωστή παρακολούθηση του συστήματος αυτού, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει ότι τελικά τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να έχουν σωστές επιδόσεις, ότι αναμένεται όχι μόνο στον τομέα της κανονικότητας και του τακτικού χαρακτήρα, αλλά και σε τομείς οι οποίοι γίνονται ακόμα πιο σημαντικοί σε όλους αυτούς τους τομείς. Αν τα κράτη-μέλη δεν παίξουν σύμφωνα με τους κανόνες και αν το ελεγκτικό συνέδριο ή εμείς εντοπίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είχαμε εντοπίσει στο παρελθόν και υποθέτουμε ότι καταθέτουμε σωστές πληροφορίες ενώ δεν ήταν τότε θα πρέπει να υπάρξουν ε, ε, πιστοτικές μάλλον διορθώσεις κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εφαρμογή του κάθε προγράμματος. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, θα επανέλθουμε. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε ενωσιακούς υπαλλήλου, ε, γιατί ε, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και αυτό θα ήταν τεράστια απέτηση για τους ενωσιακούς υπαλλήλου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα υπάρξουν και άλλες συζητήσεις ε, με εσάς στο μέλλον. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Βέλε, Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Ο εισηγητής μας ε, για την απαλλαγή του, του προϋπολογισμού ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι ο κύριος Τόιτς. Θα ήθελα λοιπόν να του δώσω το λόγο ή δεν ξέρω λέτε να το δώσω καλύτερα στον κύριο Μπέλε. Όχι. Α, εντάξει. Ο εισηγητής λέει να λάβει το λόγο γενικός γραμματέας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να κάνω ε, κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, για θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν την Επιτροπή αυτή. Είναι θέματα που είναι πολύ σημαντικά και έχουν προκύψει στους τελευταίους μήνες. Καταρχήν να πω, έχουμε συζητήσει συχνά για την ε, εργασία, για την επικοινωνία που χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την, ε, τις ευρωεκλογές ε, είχαμε 34 εκατομμύρια Ευρωπαίους, οι οποίοι προσήλθαν επιπρόσθετα στις κάλπες και αυτή τη φορά είχαμε 202 εκατομμύρια Ευρωπαίους που συμμετείχαν σε ευρωεκλογέ. Είχαμε ε, ποσοστά ε, σημαντικά ε, και στα κράτη-μέλη, ποσοστά αύξησης. Η προσέλευση των πολύ νέων ψηφοφόρων που ήταν πολύ κακή το 21% αυξήθηκε και έφτασε περίπου το 40%. Άρα δηλαδή οι προσπάθειες που κάναμε ακριβώς σε αυτό τον τομέα, νομίζω ότι οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν. Και είδαμε ότι η κοινωνία των πολιτών και αυτή συμμετείχε πολύ πιο ενεργά. Παραδείγματο χάρη είναι στο Bayern Μονάχου, ε, την Bayern München, λόγω των ευρωεκλογών, άναψε το στάδιο με χρώμα μπλε το οποίο όμως για τη Βαβαρία είναι ένα χρώμα πάρα πολύ ευαίσθητο γιατί θυμίζει το 1860. Έχουμε λοιπόν ε, πάρα πολλούς ε, που δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται και εντωμεταξύ και το σποτ ε, μας και αυτό είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι συμβάλαμε και εμείς στον να αυτή η αυξημένη προσέλευση ψηφοφόρων. Αυτά επί του θέματος. Κατά τα άλλα υπάρχουν και τα εξή ε, στοιχεία. Το 2019 για το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας περιμένουν ότι θα έχουμε 200.000 επισκέπτες. Στο TripAdvisor είναι στην 12η θέση όσον αφορά τα αξιοθέατα των Βρυξελών. Άρα καλά τα πήγε και αυτό το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ε, αυτή η θεση οσον αφορα τα αξιοθεατα των βρυξελων αρα καλα τα πηγε και αυτο το σπιτι της ευρωπαικης ιστοριας αυτη η εμπειρια για την Ευρώπη στο Ελσίνκι από το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Είχε 100.000 επισκέπτες ε, και εκεί λοιπόν από ό,τι φαίνεται ε, καλά πήγε και αυτό το project. Βεβαίως στον ε, διοικητικό τομέα κάναμε πάρα πολλά πράγματα, νέοι βοηθοί, έχουμε 1.800 συμβάσεις ε, που συνάψαμε με βοηθούς. Αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Προσπαθήσαμε να δείξουμε ευελιξία έτσι ώστε ε, οι πληρωμές προς τους βοηθούς να γίνονται δύο φορές το μήνα. Έτσι ώστε όσοι θα είχαν νέες ε, συμβάσεις να πρέπει να περιμένουν το τέλος του μήνα. 1.200 συμβάσεις ε, για τους ε, τοπικούς, ε, συν service providers, συν agents. Εξάλλου αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συζήτηση με την Επιτροπή είναι ότι η Επιτροπή επέμεινε να ασχοληθούμε και με πρώην βοηθού οι οποίοι ενδεχομένως δεν φτάνουν τα 10 χρόνια για να θεμελιώσουν συνταξιωτικά δικαιώματα. Εκτός από τρία άτομα ε, περίπου 170 βρήκαμε κάποια λύση. Αυτοί είτε συνήψαν βραχυπρόθεσμες συμβάσεις είτε προσελήφθησαν εκ νέου. Ε, για τους 170 βρέθηκε λοιπόν μια λύση για το συνταξιοδοτικό και αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει και τις προσδοκίες πολλών από το τι περιμένουν από εμάς. Καλό λοιπόν το αποτέλεσμα. Όσον αφορά το καλοκαίρι είχαμε αρκετά προβλήματα, ε, αλλάξαμε ουσιαστικά το το θέμα του Προεδρείου ε, και των γραφείων. Ε, τώρα οι βουλευτές έχουν δικό τους γραφείο στο Στρασβούργο και δεν είναι αναγκασμένοι να το μοιράζονται με τους βοηθούς τους ε, και αυτό μπορέσαμε να το πετύχουμε γιατί η διοίκηση έχασε 400 γραφεία αναδιατάξαμε ανοιχτούς χώρους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο ε, και αυτοί έκαναν κάποιες αλλαγές, δεν τους άρεσε βέβαια, αλλά εμείς επιμείναμε ότι καταρχήν οι βουλευτές πρέπει να έχουν καλές συνθήκες εργασίας. Στις Βρυξέλλες ε, για όλες τις πολιτικές ομάδες ε, έχουμε δύο γραφεία αναβουλευτή και ένα για το βοηθό. Στις Βρυξέλλες είχαμε και ουσιαστική ανακαίνιση. 2.400 ε, μονάδες ανακαινίστηκαν το καλοκαίρι και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες ε, για αυτό που έκαναν, γιατί οι συνεργάτες τουλάχιστον ε, αυτοί, οι θυγόμενοι, επέτος το καλοκαίρι δεν έκαναν διακοπές. Έχουμε και νέα έπιπλα ε, θελήσαμε να είμαστε λειτουργικοί, όχι ε, να ε, ενδώσουμε στη χλειδί και από το Νοέμβρη ε, θα είναι κάπως εξατομικευμένα τα έπιπλα, δηλαδή δεν θέλουν όλοι οι βουλευτές να έχουν σαλονάκι, άλλοι θέλουν, άλλοι δεν θέλουν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσουμε, έτσι θα εξατομικεύσουμε τον χώρο και θα έχετε έναν ηλεκτρονικό ε, κατάλογο να μπορείτε να διαλέξετε. Είδατε, μπορούμε να προσφέρουμε σαλονάκι, μπορούμε να προσφέρουμε κουζινούλα και αυτό διευκολύνει την εργασία των Ευρωβουλευτών. Ένα άλλο θέμα είναι το Brexit ε, που μας απασχολεί και διοικητικά γιατί υπάρχουν ε, κανόνες ε, οι οποίοι ε, προβλέπουν συγκεκριμένους περιορισμούς όταν τελειώνει μια θητεία. Τώρα δεν ξέρουμε θα τελειώσει η θητεία των Βρετανών βουλευτών ή όχι. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Και αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές και ενδεχομένως στις 31 Οκτωβρίου να τα ξαναπούμε, σας λέω, είμαστε πολύ ευέλικτοι γιατί οι ε, Βρετανοί ε, κάνουν τη θητεία τους με πολύ, σε πολύ δύσκολες ε, συνθήκες. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι. Και το τελευταίο που θέλω να πω, τον εκλογέν Προεδρείο, η μισή είναι καινούργοι. Στις 3 και 4 Οκτωβρίου θα έχουν αυτές τις ειδικές, μια ειδική συνεδρίαση, τα White Days που κάνουν, ε, το Προεδρείο θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα πρόγραμμα εργασίας, να συμφωνήσει για το ποιες είναι οι προτεραιότητες κατά τη διάρκεια αυτής της ε, θητείας. Και ενδεχομένως το Προεδρείο να υιοθετήσει και θέματα που υπήρχαν ήδη από το προηγούμενο Προεδρείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα. Φθινόπορο Η ή έρχεται και ξεκινά και η νέα θητεία, νέα εντολή. Και θα συναντηθούμε από ό,τι φαίνεται ε, πολλές φορές με τον Γενικό Γραμματέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ε, έκθεση και την προφορική παρουσίαση σήμερα. Θα ήθελα σύντομα να σας πω ποιος είναι ο λόγος της σημερινής αυτής ε, ανταλλαγής απόψεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας συζητήσαμε για την απαλλαγή του 2017 και λάβαμε αποφάσεις. Χορηγήσαμε απαλλαγή και διατυπώσαμε συστάσεις. Ο Γενικός Γραμματέας τώρα κάνει μια αναφορά σε ό,τι αφορά την συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις αυτές. Και έχουμε και την έκθεση απαλλαγής για το 2018. Ξεκινά λοιπόν η νέα διαδικασία. Οπότε και ε, δεκάδες ερωτήσεις ε, θα λάβετε κύριε Γενική Γραμματέα στο πλαίσιο αυτής της νέας διαδικασίας. Το θέμα είναι να δούμε ε, και να κάνουμε μία διάκριση για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, αν μιλάμε για την απαλλαγή του 17 ή αν μιλάμε για την απαλλαγή του 18. Δεν θα ήθελα τώρα εδώ να προκαταλάβω κάποια πράγματα και ούτε θέλω να μιλήσω για το 2018, δεν θέλω να προτρέξω. Δύο πράγματα έχω να πω. Το πρώτο, Δεν ξέρω κατά πόσο να είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Όχι ότι θέλω να εκφράσω παράπονα και δυσαρέσκεια, αλλά... Έχουμε το θέμα της ε, φιδωλής ε, χρήσης των ε, φορολογουμένων. Έχουμε το νέο ταξιδιωτικό γραφείο, πριν είχαμε ένα άλλο, υπήρξε διαδικασία διαγωνισμού. σε ό,τι αφορά αυτό το νέο ταξιδιωτικό γραφείο, δεν άκουσα και το λέω έτσι διπλωματικά καμία θετική κριτική από κανέναν. Πώς είναι δυνατόν να κοστίζουν ε, ε, οι ίδιες ουσιαστικά υπηρεσίες ε, το ίδιο, μάλλον περισσότερο μέσα στο κοινοβούλιο από ότι εκτός κοινοβούλιο. Γιατί να πρέπει εμείς να πληρώνουμε περισσότερο για τις ίδιες υπηρεσίες. Εδώ πρόκειται πάντα για χρήματα φορολογμένων. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Δεν είναι δυνατόν να δαπάνουμε περισσότερα για την ίδια υπηρεσία Ιδίω όταν στην ε, αγορά δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια αύξηση των τιμών. Έχετε εσεί ε, κάποια εξήγηση. Ήταν πιο αποδοτικό ό,τι αφορά τη χρήση των ε, χρημάτων φορολογουμένων. το προηγούμενο εξωτικό γραφείο είναι αυτό. Και ένα θέμα που πάντα έρχεται και ξανάρχεται είναι το δεύτερο που θέλω να θέσω. Μεγάλωσα στην Ουγγαρία, σε μια ε, σχεδιαζόμενη οικονομία, προγραμματισμένη και δεν υπήρχε ελεύθερη αγορά, δεν υπήρχε ελεύθερος ανταγωνισμός, αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι όλα τα ξενοδοχεία στο Στρασβούργο ξέρουν επακριβώς πότε συνεδριάζει το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Και τριπλασιάζεται η τιμή του κάθε δωματίου ξενοδοχείου τις μέρες ε, της Ολομέλειας και μετά ξαναπέφτει ναι, εντάξει, μπορεί να παίζουν ε, ρόλο κάποια κριτήρια, ότι είναι κάποιες ημερομηνίε φίξ ε, και τα λοιπά. Όμως οι συνεργάτες ε, του Κοινοβουλίου, άλλοι που έρχονται στο Κοινοβούλιο, για αυτούς πληρώνουν φορολογούμενους ουσιαστικά τη διαμονή τους, τα οδηπορικά τους. Δηλαδή να κοστίζει ένα δωμάτιο ξενοδοχείο 80 και να κοστίσει 200 ευρώ στην ε, Ολομέλεια, κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Φυσικά και σεβόμαστε την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό. Όμως παρακαλώ, πρέπει να το έχετε και αυτό υπόψη, να δούμε μήπως μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα για να αποτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα. Να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί δηλαδή στη χρήση των κονδυλίων, γιατί πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων. Δεν θέλω να στραφώ ενάντια στους ε, ιδιοκτήτες των, ή τους ε, διαχειριστές των ξενοδοχείων, αλλά αν πάω στη Γερμανία, ε, εκεί δεν βλέπω αντίστοιχα φαινόμενα σχροκέρδειας. Να δώσουμε το λόγο στον Γενικό Γραμματέα. Ο εισηγητή ε, επισήμανε ότι υπάρχουν ε, θέματα που έρχονται και επανέρχονται. Αυτό είναι αλήθεια. Το ταξιδιωτικό γραφείο καταρχήν είναι το Carlson Wagon Lee. Είχαμε συνεργαστεί με αυτούς ε, και κατά το παρελθόν σε αυτή τη νέα διαδικασία του διαγωνισμού ε, αποφασίσαμε να ε, επιβάλλουμε και άλλε προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη ανοιχτή το μεσημέρι, παλιά δεν ήταν. Ή ε, το θέμα των εισιτηρίων ε, να μπορεί κανείς να κάνει καθάριση εταιρείου χωρίς ε, χαρτί και ε, υποστήριξη 24 ώρη. Παρ' όλα αυτά βέβαια όταν αλλάζει το πρακτορείο Προφανώς ε, προκύπτουν δυσκολίες, ε, μερικοί συνεργάτες είναι ίδιοι, άλλοι είναι καινούργοι, πρέπει και αυτοί να συνηθίσουν, αλλά ακόμα και αν είναι οι ίδιοι που δούλευαν μέχρι τώρα για μας, πρέπει και αυτοί να εργαστούν με ένα νέο ε, σύστημα πληροφορικής. Υπήρξε βέβαια κάποια εκπαίδευση το Δεκέμβρη, παρόλα αυτά όμως τα προβλήματα προκύπτουν στην πράξη και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα ε, που μας ε, απασχολούν. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι το ποσοστό των διαμαρτυριών και της ε, έλλειψης ικανοποίηση, αυτό το ποσοστό παραμένει το ίδιο 0,04% των συναλλαγών. Άρα δηλαδή δεν διαπιστώσαμε ότι σε σχέση με τον προηγούμενο πάροχο ότι έχει προκύψει κάποια επιδείνωση. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που το θίξατε κι εσείς, δηλαδή όλο και περισσότεροι ε, ταξιδιωτικοί πράκτορες ε, ε, κάνουν και απευθείας πωλήσει, δηλαδή ε, πολλοί ακυρώνουν τον ε, μεσάζοντα, κάνουν καλύτερες προσφορές και γι' αυτό και εγώ πολύ συχνά βρίσκω τιμές ε, που είναι πιο ευνοϊκές. Μερικές φορές αυτό σχετίζεται με το τι είδου εισιτήριο είναι. Ε, το θέμα, παραδείγματο χάρη, της ακύρωσης, δυνατότητα ακύρωσης. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πολλές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες απευθύνονται κατευθείαν στην αγορά και έτσι γλιτώνουν τα χρήματα για τους μεσάζοντες. Όσον αφορά την κατάσταση των ξενοδοχείων στο Στρασβούργο, θέλω να σας πω ότι γενικά όσον αφορά τον, την ποσότητα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ε, ξενοδοχείων στο ε, Στρασβούργο. Ίσως βέβαια να αυξήθηκε και η ζήτηση. Ε, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα με τις τιμές ξενοδοχείων στο Στρασβούργο παραμένει είναι ξεκάθαρα θέμα αγοράς. Αυξάνεται η προσφορά, αλλά αυξάνεται και η ζήτηση, δυστυχώς, ε, για την εβδομάδα της Ολομέλειάς μας. Το έχουμε συζητήσει με τις αρχές του Στρασβούργου εδώ και κάποια χρόνια. Συναντιόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο αρμόδιος αντιπρόεδρος ε, συναντιέται με τις αρχές του Στρασβούργου και οι αρχές του Στρασβούργου ε, δεσμεύτηκαν να φτιάξουν μια μελέτη μελέτη σκοπιμότητας. Ε, να ε, υπάρχει ενδεχομένως αγορά ε, δωματίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά αυτά να διατίθεται στους ενδιαφερόμενους. Έτσι ίσως θα πέσουν οι τιμές και κάνουμε κάποιες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που τέτσαν και τώρα πάω στους ε, σκιοδησηγητές η κυρία Γκραπίνη από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα και να τον καλωσορίσω κιόλας Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που σήμερα ακούμε νέα καλά. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική περίοδος αυτή που διανύουμε και νομίζω έχετε παρουσιάσει κάποιες από τις θετικές εξελίξεις. Ο συνάδελφος εισηγητής έθεσε ορισμένα θέματα τα οποία και εγώ θα ήθελα να θέσω. Ίσως θα μπορέσετε να απαντήσετε όμως και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής. Θα ξεκινήσω χαιρετίζοντας το ότι η Γενική Γραμματεία είναι πιο ισόρροπη σε επίπεδο φίλων. Αυτό με ικανοποιεί. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον, να διαπιστήσουμε ότι η ισορροπία των φίλων είναι σε καλύτερη φάση σήμερα και θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος των γυναικών στο Κοινοβούλιο. Μιλήσατε επίσης και για τον εξυγχρονισμό αλλά δεν μιλήσατε για μία μορφή εξυγχρονισμού πολύ σημαντική, την σελίδα web του Κοινοβουλίου. Ε, σκοπεύετε να ανανεώσετε, να εξυγχρονίσετε την ε, ιστοσελίδα αυτή, γιατί την έχουμε ανάγκη και πρέπει να ανανεωθεί. Έχετε κάποιες ιδέες έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να τον εξυγχρονίσουμε ε, την ιστοσελίδα αυτή. Αναφερθήκατε και στις διαδικασίες προσλήψεων. Γνωρίζετε ότι η προηγούμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή είχε ζητήσει να υπάρξει ένα εγχειρίδιο ε, για οδηγιών για τους υπευθύνου πληρωμών. Θα πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι πληρωμών, όλοι οι διατάκτες ε, να γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα πράγματα για να αποφεύγουμε ε, κάποιες συγχύσεις και ελλείψεις αντιστοιχίας. Τώρα για τους λεγόμενους σταζιέρ. Μιλήσατε για τους βουλευτές, για τους συνεργάτες, αλλά έχουμε και τους ταζιέρ, οι οποίοι εργάζονται για μας. Η πολιτική μου ομάδα λοιπόν εδώ είναι ανήσυχη. Ε, θα μπορούσαν να πληρώνονται με προκαταβολή η σταζιέρα αυτή. Μια άλλη ερώτηση για τα γεύματα. Έχουν κάποιες δυνατότητες στην κατίνα, αλλά μόνο κατά ένα ποσοστό του μισθού τους. Βλέπουμε επίσης ότι οι τιμές στα εστιατόρια έχουν αυξηθεί πολύ, ενώ η ποικιλία δεν έχει αλλάξει ε, λοιπόν, σκεφτείτε όχι μόνο το, την ευκολία, αλλά και τους οικονομικούς όρους. Αν για το ίδιο φαγητό πρέπει να πληρώνουμε περισσότερα, τουλάχιστον να πρέπει να είχαμε καλύτερη ποιότητα. Και κάτι το οποίο επίσης έχει μεγάλη σημασία είναι το θέμα της ασφάλειας. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονες στην διάθεσή σας θα μπορούσατε παρακαλώ κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής εντολής να υπάρξει ε, μια σωστή ενημέρωση ε, για την ασφάλεια στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Ε, για τα θέματα του γραφείου ταξιδίων δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα είπε ο συνάδελφος. Υπάρχει ένα κοινωνικού χαρακτήρα θέμα, μιας και προέρχομαι από την ομάδα των σοσιαλιστών. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ ε, τα προβλήματα των ευρωβουλευτών γυναικών που είναι μητέρες και θέλουν να αφήσουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό αλλά δεν είναι δυνατό να το κάνουν με τα οχήματα του Κοινοβουλίου. Μπορείτε να δώσετε την δυνατότητα αυτή στις γυναίκες μητέρες συναδέλφους. Αυτό θα ήταν κάτι που θα εκτιμήσουμε δεόντως. Τώρα, η διακοπή των συμβάσεων για τους ε, επιστοποιημένους και τοπικούς συνεργάτες. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από το επίδομα ανεργίας. Και αυτό είναι, ισχύει και για την ιατρική τους ε, ε, πρόνοια, η ασφάλεια. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ προσεκτική, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τους σεβαστείτε λίγο περισσότερο από ό,τι το κάνετε και θέλω να σας ευχαριστήσω και για όλες τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε μέχρι τώρα. Ω σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας των σοσιαλιστών είμαι πεπισμένη ότι σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής κάποια από τα προβλήματα θα τα λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκραπίνη που είστε και εισηγήτρια για το 18 η σκιώδης. Επόμενος, η επόμενη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γενικό Γραμματέα για την παρουσία του εδώ και για την έκθεσή του. Η συζήτησή μας αφορά την απαλλαγή για τον 2017 ουσιαστικά. Ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά μακριά στον χρόνο, διότι εγώ είμαι νέος εδώ θα είχα και εγώ πολλές ερωτήσεις να σας θέσω για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα. Και ως κοσμήτορ ε, είχα ήδη την δυνατότητα να σας θέσω αρκετές ερωτήσεις ε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Προεδρείου. Ε, το θέμα σήμερα λοιπόν είναι η απαλλαγή για το 2017. Οι ερωτήσεις τις οποίες έχασαν οι συναδελφοί επανέρχονται συστηματικά στις ερωτήσεις τις οποίες ε, θέτουν οι βουλευτές τους κοσμήτορες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φρόιντε, είστε σκιώδη εκ μέρου των Πρασίνων. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέλε, που είστε εδώ. Έχω και εγώ ναι, λίγες ε, ερωτήσεις ε, που ε, επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και κάποιες καινούργια σε ό,τι αφορά την αποζημίωση του κόστους. Εδώ και κάποιο καιρό αλλάξαμε στην προηγούμενη θητεία το καθεστώς, αλλάξαμε τους κανόνες και μου είπαν να τα καταγράφω όλα αυτά σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι και ε, υποχρεωτικό να μπαίνει αυτή η αποζημίωση εξόδων σε διαφορετικό λογαριασμό. Υπάρχει πράγματι όμως αυτός ο ξεχωριστός λογαριασμός ε, από τους συναδέλφους ε, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτή την αποζημίωση έχουν όλοι οι συνάδελφοι ήδη φτιάξει ειδικό λογαριασμό και υπάρχει κάποιος ελεγκτής που ελέγχει τα παραστατικά από καιρούς καιρών. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ε, θελοντικό σταξιδοτικό ταμείο, ε, από ό,τι ξέρω, κάποια στιγμή το Προεδρείο ε, αποφάσισε το Δεκέμβριο του 2018 Ε, να μην ασχοληθεί τόσο πολύ με το τι θα γίνεται με τα προβλήματα ε, αυτά. Όμως δεν θέλουμε τα πράγματα να γίνουν ακόμα χειρότερα ε, σε ό,τι αφορά το ταμείο αυτό. Εξάλλου ξέρουμε ότι οι βουλευτές ε, παίρνουν ήδη πολύ καλές αμοιβέ και δεν θα ήθελα να φαίνεται από να βλέπουν ότι σου θα εξασφαλίσουν πάρα πολλά περισσότερα. Επίσης, τα δύο τρίτα ε, των ε, βουλευτών είμαστε νέοι βουλευτές. την προηγούμενη θητεία άλλαξε και ο στερικός κανονισμός ε, σε ό,τι αφορά τις ε, ε, δηλώσεις των βουλευτών για το, τα άλλες δραστηριότητες, άλλα επιτιδεύματα που θα δηλώνονται μόνο εδώ. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει κάτι. Υπενθυμίσατε στους βουλευτές ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση δυνάμη του κανονισμού πλέον Και τι γίνεται με τους βουλευτές που έφυγαν. Υπάρχει ενδεχομένως ε, κάποιος που μπορεί να θέλει να εργαστεί σε έναν ε, δημόσιο φορέα. Υπάρχει θέμα σύγκρουση συμφερόντων και τι γίνεται. Ξέρει το κοινοβούλιο ποια είναι η νέα ασχολία των προηγούμενων βουλευτών ή συνεργατών. Και τι κάνετε, με κάποιο τρόπο υπάρχει η δυνατότητα ή η υποχρέωση να το δηλώσουν για να μπορεί κανείς να διαπιστώνει πού μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Και η τελευταία ερώτηση που έχω έχει να κάνει με κάτι που συζητήσαμε σήμερα το πρωί, την απαλλαγή για την ΙΑΣΟ που για ακόμα μία φορά δεν τη χορηγήσαμε. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη Ασύλου, ΕΑΣΟ. Ένα από τα μέλη ε, του, της διοίκησης ε, ε, είναι σε διαθεσιμότητα ή τέλος πάντων υπάρχει κάποια ε, διαδικασία σε βάρος του, κατηγορίες για κακοδιαχείριση σε βάρος του κτλ. Αυτός όμως ο υπάλληλος Νομίζω ότι είναι πλέον εδώ ε, ε, υπάλληλο στο Κοινοβούλιο ε, και θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον ισχύει αυτό ή όχι. Είναι δυνατόν άνθρωποι για τους οποίους έχει κινηθεί τέτοια διαδικασία να μπορούν να ανακυκλώνονται μέσα στη, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να μην λογοδοτούν για αυτά που έχουν κάνει κάπου αλλού. Ίσως να ακούσουμε μία απάντηση ενδιαμέσως από τον Γενικό Γραμματέα, γιατί είναι πολλές ε, ερωτήσεις. Ε, μην τις ξεχάσετε και θα συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν όσον αφορά τα θέματα που έθεσε η κυρία Γκραπίνη για το θέμα του φίλου, της διάστασης του φίλου πράγματι νομίζω ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση. Όταν εγώ ανέλαβα το αξίωμά μου είχαμε μία ε, μάλλον με συγχωρείτε, 21% ε, ήταν γυναίκες, τώρα είναι το 40% γυναίκες στα στελέχη. Άρα δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμό. Και αυτό σημαίνει ότι κατ' ουσίαν τον τελευταίο καιρό ε, έχουμε διορίσει περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να φτάσουμε να εξηγήσουμε αυτό το ποσοστό. Κάτι γίνεται λοιπόν. Όσον αφορά τις ε, διευθύντριες, ε, το 37% είναι γυναίκες. Όταν τελείωσε η θητεία ήταν 35%, άρα και εκεί βελτίωση. Και στο επίπεδο των τμήματαρχών, εκεί μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση μέχρι το τέλος της θητείας μπορούμε να έχουμε 50% ε, γυναίκες σε επίπεδο τμήματαρχών. Βέβαια, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις που θα λάβει το Προεδρείο, γιατί εκείνο διορίζει. Ε, προφανώς, ε, στο επίπεδο γενικών διευθυντών, εκεί φύγανε αρκετές γυναίκες και βέβαια αυτές δεν αντικαταστάθηκαν απαραίτητα από γυναίκες. Εκεί δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Εγώ προσωπικά έλαβε την απόφαση στην ε, Επιτροπή για Ανώτερα Στελέχη να ε, διορίσουμε μία ε, δεύτερη Γενική Διευθύντρια ως μόνιμο μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου για να διασφαλίσουμε ικανοποιητική εκπροσώπηση και να μην είναι γυναίκες πάντα σε θέση μειοψηφίας. Όσον αφορά την ιστοσελίδα, πράγματι έχουμε μια τεράστια ιστοσελίδα και ακριβώ γιατί είναι τόσο μεγάλη και με πολλές λεπτομέρειες είναι δύσκολο να ψάξει κανείς κάτι στην ιστοσελίδα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι και στην αναζήτηση ε, με τη μηχανή Google. Εκεί τα πάμε πολύ καλύτερα. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία τα πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Αν γράψει κανείς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, δεν πάει απαραίτητα στην τρίτη τέταρτη θέση, πολλές φορές πάει στην πρώτη θέση και εξαρτάται βέβαια πολλές φορές από το πώς ακριβώς ε, έχουν ε, οριστεί αυτές οι στοσελίδες. Ίσως και εκεί μπορούμε να επιτύχουμε μια βελτίωση. Αλλά με την αρχή της νέας θητείας καταβάλλονται προσπάθειες να βελτιωθούμε και στον τομέα αυτό. Ε, όσον αφορά το να υπάρχουν πληροφορίες για τις νέες θέσεις, αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Πρακτική βέβαια δυσκολία είναι ότι έχουμε 28 διαφορετικά νομικά συστήματα που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια θέματα για τους ε, επιτόπιους ε, βοηθούς που είναι κοινά αλλά και πάρα πολλά άλλα που είναι διαφορετικά. Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε γιατί υπάρχουν όρια Βεβαίως ε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Στους ε, εκπαιδευόμενους, στους ε, σταζιέρ, στο Προεδρείο, εκεί έχουμε αποφασίσει για νέους κανόνες και αυτοί θα λαμβάνουν προκαταβολή για το ταξίδι όπως και η βοηθή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους σταζιέρ γιατί δεν έχουν πολλά χρήματα και για τους σταζιέρ εξακολουθούμε να έχουμε ένα επίδομα για να μπορούν να φάνε στην καντίνα ε, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και συζητάμε ακόμα με τους ε, παρόχους ε, της καντίνας, κατά πόσον μπορούμε ε, να έχουμε και μεγαλύτερη και καλύτερη βελτίωση. Όσον αφορά στην ασφάλεια, νομίζω ότι κάναμε πάρα πολλά, κυρίως όσον αφορά τη σωματική ασφάλεια. Για το διαδραστικό app πρέπει να το ελέγξουμε. Εγώ προσωπικά είμαι λιγάκι επιφυλακτικός όσον αφορά τις δυνατότητές μας. Το να έχουμε ένα απόλυτα ασφαλές ε, μια τέτοια εφαρμογή, δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε. Ε, όσον αφορά τώρα τους οδηγούς, ε, ε, οι οδηγοί δεν μπορούν να κάνουν ενδιάμεσες, να σταματάνε ενδιάμεσα, όμως οι κοσμήτορες το συζητάνε και το θέμα θα επανέλθει στις συνεδρίες του Οκτωβρίου. Δεν έχει κλείσει το θέμα αυτό και έχοντας κατά νου ότι οι κοσμήτορες θα το ξανά συζητήσουν, βλέπετε ότι το θέμα το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Και ε, αυτό ε, πράγματι το έχουμε κατανοήσει ως πρόβλημα. Τώρα, εάν ε, για πρώην συνεργάτες υπάρχουν συγκεκριμένες συγκεκριμένα προβλήματα να μου τα πείτε. Ο κύριος Φρόιντ ε, έθεσε ερωτήματα που αφορούν καταρχήν ε, στην ε, αποζημίωση κόστους. Δεν έχουμε στοιχεία για το... Δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα για το πώς οι βουλευτές έχουν αποκτήσει ειδικό λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό. Δεν έχουμε τέτοια στατιστικά δεδομένα. Ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά αν σας ενδιαφέρει να το ψάξουμε και να δούμε. Ε, το, η αποζημίωση, η γενική αποζημίωση δαπανών, αυτή η συζήτηση έγινε στο Προεδρείο, παρέμεινε ένα καταποκοπή ποσό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει εκαθάριση. Ως εκ τούτου έχουμε ακόμα το παλιό σύστημα, βέβαια με κάποιες αλλαγές και ως εκ τούτου θα υπάρχει διαφάνεια. Για το συνταξιοδοτικό ταμείο, το Προεδρείο μετά από δική μου πρόταση ε, έλαβε δύο μέτρα. Πρώτον, την αύξηση ε, του ορίου συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 έτη. Και δεύτερον, να προβλέπετε ειδική σφορά της τάξης του 5% που πρέπει να καταβάλουν οι συνταξιοδοτούμενοι. Και τα δύο αυτά μέτρα ε, βέβαια αμφισβητούνται αυτή τη στιγμή ε, διότι έχουν προσφύγει πρώην ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εξετάζεται το κατά πόσο το Κοινοβούλιο είχε το δικαίωμα να προβεί σε αυτήν την αλλαγή πριν από 10 χρόνια είχαμε κάτι παρεμφερές και το δικαστήριο αποφάνθηκε τότε ε, το δικαστήριο επιβεβαίωσε όλες τις αποφάσεις του Προεδρείου ως σωστές και αναλογικές. Το κατά πόσον θα ξαναγίνει αυτό θα το δούμε. Την τελευταία φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας ε, επιβεβαίωσε ότι κατ' ουσίαν πρόκειται για επικουρική σύνταξη και δεν πρόκειται για την κύρια σύνταξη και επιπλέον ε, δεν αφορά το σύνολο της ε, θητείας. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τέτοια περικοπή υπηρεσιών, παροχών. Το θέμα είναι πού βρίσκεται το όριο. Αυτό το εξέτασε η δική μας η νομική υπηρεσία και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουμε εξαντλήσει τα όρια ή κατά πόσον υπάρχει ακόμα κάποιο περιθώριο ή μήπως έχουμε ξεπεράσει το όριο. Τη στιγμή λοιπόν που θα έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και για αυτά τα μέτρα θα μπορούμε να υπολογίσουμε καλύτερα το κατά πόσον έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας, αν έχουμε ακόμα κάποιο περιθώριο και ενδεχομένως κατά πόσον μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα από το Προεδρείο που θα περιορίζει την επιβάρυνση για το φορολογούμενο ή ενδεχομένως να δούμε μήπως έχουμε ξεπεράσει τις δυνατότητες μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην περίπτωση αυτή τα μέτρα που έχουμε λάβει καταπίπτουν. Ε, η απόφαση του δικαστηρίου θα μας δώσει ένα προσανατολισμό να δούμε τι θα κάνουμε, αν θα προχωρήσουμε περισσότερο ή μήπως έχουμε εξαντλήσει ήδη πλήρως τις ε, νομικές μας δυνατότητες και θεωρώ ότι όταν θα υποβληθεί η απόφαση του δικαστηρίου, το Προεδρείο θα εξετάσει εκ νέου αυτό το θέμα για να δει κατά πόσο μπορεί να λάβει και άλλα μέτρα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία θα λαμβάνεται ένα συγκεκριμένο μέτρο, παραδείγματο χάρη το πάγωμα των παροχών. Αυτή είναι η τρίτη εναλλακτική λύση που υποβλήθηκε στο Προεδρείο. Ακόμα λοιπόν και αν προέκυπτε και αποφασιζόταν των παροχών, ε, το έλλειμμα του συνταξιωτικού ταμείου αυτή τη στιγμή επουδενή δεν θα καλύπτεται. Όμως ε, το Κοινοβούλιο με την θέση σε ισχύ του ε, καταστατικού βουλευτών ανέλαβε κάποιες υποχρεώσεις έναντι του συνταξιωτικού ταμείου. Αυτά από το 2009 όπου δεν υπήρχε κοινή ε, υπηρεσία που να προσφέρεται κοινή παροχή σε όλους τους ευρωβουλευτές, μόνο εθνική παροχή. Το 2009 λοιπόν άλλαξαν τα πράγματα με αυτήν την απόφαση θα δούμε τι θα κάνουμε. πάση περιπτώσει θα, παρα... θα εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα και επειδή το Κοινοβούλιο ευθύνεται για αυτό το έλλειμμα, ε, αυτό το έλλειμμα εντάσσεται στον προεπολογισμό του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον αυτή είναι η αξιολόγηση της νομικής μας υπηρεσίας. Για την ε, πλήρη απασχόληση των συνεργατών μας. Υπάρχουν διάφορα συστήματα, διάφορες δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι πρώην στελέχη μας, οι οποίοι έχουν μία περίοδο όπως θα την χαρακτηρίζει cooling off. Βέβαια δεν έχουμε εκεί αυτή τη στιγμή κανένα και δεν ζήτησε κανείς ε, να προσληφθεί εκ νέου. Κατά κανόνα, οι συνεργάτες μας απασχολούνται μέχρι τη συνταξιδότησή τους. Έχουμε βέβαια την ειδική περίπτωση των βοηθών. Οι βοηθοί, αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, οφείλουν να την κοινοποιήσουν. Άρα δηλαδή και εμείς ε, ε, δεν είμαστε σε θέση όπου να ελέγχουμε πού ακριβώς απασχολείται ο καθένας. Αλλά αν τελικά κάποιος κάνει κάποια δουλειά που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων, τότε οι βοηθοί θα πρέπει να το δηλώσουν. Έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις όπου πράγματι έγινε μια τέτοια δήλωση που εξετάστηκε ε, και θυμάμαι μία περίπτωση ή κάποιες περιπτώσεις όπου ε, αρνηθήκαμε απασχόληση σε βοηθούς ε, γιατί υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων με την τρέχουσα απασχόληση ή θα προέκυπτε σύγκρουση συμφερόντων. Όσον αφορά τώρα συνεργάτες μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο θέμα της χορήγησης ασύλου, αυτό είναι θέμα καταστατικού. Αν κάποιος είναι υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως ε, είχε κάποια μερική απασχόληση σε κάποιο άλλο θεσμό, προφανώς και έχει το δικαίωμα να επανέλθει στην πρώην απασχόλησή του. Βέβαια ε, θα πρέπει κανείς να εξετάσει το κατά πόσον ε, υπήρξαν ποινικά κολάσιμες πράξεις ε, κατά την προηγούμενη εργασία του, αλλά ξέρετε αν έχει αν υπάρχουν κάποιες υποψίες για ποινικά κολάσιμες πράξεις, κανείς δεν μπορεί να απολυθεί. όλοι επανέρχονται στην απασχόλησή τους στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν υπήρξαν ε, πειθαρχικές ε, παραβάσεις, ε, αυτές εξετάζονται και διώκονται ή όχι ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας. Ξέρω ότι στην ΕΑΖΟ υπάρχουν πάρα πολλές πειθαρχικές διαδικασίες και όσο τρέχουν αυτές οι διαδικασίες. Δεν μπορεί κανείς να απολύσει κάποιον, ο συνάδελφος κύριος Φρόιντ. Κοιτάξτε, όσον αφορά α, τους βοηθούς οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά από την αποχώρηση κάποιων ευρωβουλευτών που δεν επανεξελέγησαν. Δεν ξέρω, τι, δεν το γνωρίζω αυτό. Το ρωτάω γιατί με βάση το καταστατικό ως τροποποιήθηκε από το 2008 αναφέρεται στο καταστατικό του Κοινοβουλίου ότι ε, τη δουλειά που κάνει κανείς μετά την απασχόληση σε ένα ευρωβουλευτή πρέπει να τη δηλώνει. Κοιτάξτε, το θέμα είναι κατά πόσον το δηλώνουν οι ίδιοι ευρωβουλευτές ή κατά πόσον θα πρέπει να το ελέγχει η διοίκηση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θα το ελέγξω. συνάδελφος ε, Τσε. Καταρίνα Τσε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. General for, uh, being with us. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέλερ. Ως νέο μέλος θα ήθελα να θέσω ορισμένα θέματα στα οποία θα έλεγα μου χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Κάθε μήνα πηγαίνει το κοινοβούλιο εκεί και πηγαίνουν τα αυτοκίνητα για να μας εξυπηρετούν εκεί με ένα οδηγό. Το υπόλοιπο προσωπικό που πηγαίνει στο Στρασβούργο δεν έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα αυτοκίνητα του Κοινοβουλίου, τα οποία πηγαίνουν άδεια. Εδώ παρακαλώ χρειάζομαι μία αλλαγή, μία τροποποίηση του κανονισμού, έτσι ώστε θα γλιτώσουμε και χρήματα, θα γλιτώσουμε φυσικά και το ίχνος μας το περιβαλλοντικό, το οποίο είναι βασική προτεραιότητα για μας εφόσον δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα την άποψή σας αν κάτι τέτοιο λοιπόν είναι εφικτό. Η δεύτερη ερώτηση. If I'm correct in the... Α, τα γενικά έξοδα, την αποζημίωση γενικών εξόδων. Ε, είχε υπάρξει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εντολής μια ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Έχετε δημιουργήσει και στο νέο Προεδρείο. Υπήρχε μια διαφορά ανάμεσα στην Ολομέλεια ίσως και το, και το Προεδρείο γι' αυτό. Καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, τρίτη ερώτηση. Έμαθα ότι υπάρχει ε, δυνατότητα ε, για εθελοντική, αν θέλετε, συνεισφορά σε επίπεδο νομοθετικό. Ε, θα ήθελα να μάθω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ποιοι την έχουν χρησιμοποιήσει και καλό θα ήταν να οι πληροφορίε αυτές κυκλοφορούσαν περισσότερο έτσι ώστε όλοι να συνειδητοποιούν ακριβώς τι δυνατότητες υπάρχουν έτσι ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Και μια τέταρτη ερώτηση, τελευταία. Όταν α, εμείς τεκμηριώνουμε τα εσωτερικά μας ταξίδια στις χώρες μας, λέμε σε ποιο μέρος πάμε και τον αριθμό του αυτοκινήτου. Προσωπικά, μερικές φορές είναι περίεργα γενναιόδοροι οι υπολογισμοί τους οποίους κάνει το Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα ήθελα να βρείτε ένα κάπως πιο διαφανές σύστημα και έτσι να εξοικονομήσει χρήματα το Κοινοβούλιο και οι φορολογούμενοι. Ε, <clears throat> um, Ευχαριστώ τον κύριο Βέλε για μια ακόμη φορά τρία σημεία τα δύο είναι σημεία κριτικής και ε, το τρίτο είναι θα έλεγα εκθεαστικό για τον κύριο Βέλε. Θα το αφήσω τελευταίο όμως για να μας μείνει μια καλή επίγευση. Ε, θα ήθελα να ακούσετε παρακαλώ τις δύο πρώτες παρατηρήσεις προσεκτικά. Είναι πολύ συγκεκριμένα θέματα. Θεωρώ ότι πολλές φορές είμαστε λίγο γενικόλογοι. Συχνά είμαστε πολύ γενικόλογοι. Ενώ αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην καθημερινότητα του Κοινοβουλίου. Πρέπει να γλιτώσουμε χρήματα και χρήματα του φορολογού. Δε πρώτο είναι τα υπηρεσιακά οχήματα. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε προσοχή σε αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες δίδονται από την υπηρεσία στους οδηγούς. Εδώ και έξι μήνες περίπου, ίσως και παραπάνω. Λέγεται με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο ότι αν το μέλος μέσα σε πέντε λεπτά δεν εμφανίζεται το σημείο και την ώρα συνάντησης, τότε ο οδηγός θα πρέπει να αποχωρεί. Και φυσικά οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής λοιπόν. Αυτό είναι πραγματικά περιττό. Γιατί είναι πάρα πολύ συχνό για πρακτικούς λόγους να μην είμαστε ικανοί να είμαστε εκεί μέσα στο πεντάλεπτο. Πολλές φορές είναι 6 λεπτά, 7 λεπτά ή 8 λεπτά. Παράδειγμα. Είχαμε απέναντι τον πρόεδρο και τον υπουργό και απευθύνεται σε μένα και ξαφνικά εγώ θα σηκωθώ και θα σηκωθώ να φύγω λέγοντας ότι το αυτοκίνητο του κοινοβουλίου δεν θα περιμένει. Μα έγινε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκα έξω, δεν υπήρχε αυτοκίνητο, πήρα την υπηρεσία και του ζήτησα να επανέλθει. Ε, παίζουμε τώρα. Δεν είναι δυνατό να πηγαίνω ερχόμαστε μέσα στην πόλη. Ε, λόγω αυτού του συγκεκριμένου κανόνα, ο οποίος πρέπει να γίνει πιο ευέλικτος. Λοιπόν, παρακαλώ, σας ζητώ να το λάβετε υπόψη. Οι οδηγοί δεν είναι βλάκες, είναι καλοί επαγγελματίες και μπορούν να κρίνουν ανάλογα με την κατάσταση να μην κοιτούν συνέχεια το ρολόι και ε, λέγουν ότι αν δεν φύγουν στο πεντάλεπτο θα τους κυνηγήσει ο, επι, το, ο επόπτης τους. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Υπάρχει μια αυτόματη επιστροφή εξόδων ταξιδίων εδώ και λίγους μήνες. Ξέρω ότι είναι σε αρχική φάση ακόμα, αλλά είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη σαχλαμάρα. Όλα κολλάνε, όλα συγχέονται, γι' αυτό παρακαλώ να το ελέγξετε. Και παρακαλώ να μην εισάγετε νέα αυτοματοποιημένα συστήματα πριν σε επίπεδο πληροφορικής δεν είμαστε απόλυτα συγχρονισμένοι γιατί αυτό προκαλεί απώλεια χρόνου, προκαλεί πονοκέφαλο και όλοι νιώθουν μια βαριά δυστημία. Μέλη όπως και εγώ σύμφωνα με τη γυναίκα μου κάνομαι, κάθομαι πάρα πολύ συχνά στην πίσω σειρά είστε μια μαύρη μεσεντές και δεν αντέχω, δεν ξέρω αν είναι ότι είναι κακομαθημένος. Λοιπόν, όπως είπαμε, η αλλαγή των κανόνων αυτή είναι μια τεράστια προσπάθεια ε, για τα γραφεία και όταν γυρίσαμε ήταν θαύμα το αποτέλεσμα. 11.000 μετακινήθηκαν και όλοι πήραν τους χώρους οι οποίοι ε, τους αναλογούσαν και αυτοί οι οποίοι το πέτυχαν αυτό ε, πρέπει να τους συγχαρούμε με τον δυνατότερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πέτρη. Μια παρατήρηση και κάτι άλλο να πω για τα ταξίδια μετά. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν λογικό μετά από τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό ταμείο Εμένα δεν με αφορά βέβαια. Ίσως να ακούγαμε όμως ε, από αυτούς τους συναδέλφους που τους αφορά και που λένε ότι δεν έχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου επικουρική σύνταξη. Οπότε καλό θα ήταν ίσως να γίνει μια ανάλυση ε, του συστήματος που ίσχυε πριν από το 2009 ε, για τα δικαιώματα τα οποία έχουν μέχρι τότε στη χώρα τους. Να δούμε αν είναι για όλους επικουρικό, για άλλους δεν είναι, γιατί προς το παρόν ε, δεν έχουμε βεβαιότητα για το τι ισχύει. Καλό θα ήταν ίσως να γίνει μια τέτοια μελέτη, μια τέτοια ανάλυση για να μας ε, διαφωτίσει και εμάς ε, και να καταλάβουμε τι ισχύει. Σε σχέση τώρα με αυτά που είπε ο Πέτρη Σαρβάμα, για το σύστημα πληροφορικής Ουσιαστικά η διοίκηση είχε αυτό το καθήκον πριν και τώρα το έχουν αναλάβει οι βουλευτές. που μας ε, έχει μετακυλήσει η διοίκηση, δηλαδή ένα ακόμη βάρος. Ε, το πρόβλημα είναι γιατί να περιμένουμε και 6 φορές παραπάνω. Δεν ήταν και τόσο μεγάλο ο φόρτο για τη δίκη. Περιμένουν 8 με 12 εβδομάδες τώρα οι βουλευτέ για την αποζημίωση και αυτό δημιουργεί κάποια δυσφορία στους βουλευτέ. Βέβαια, απ' την άλλη, αν τους το ξανά στη διοίκηση και είναι ακόμα μεγαλύτερο το διοικητικό άκθος που έχουν, ίσως να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πληρωμές μας και για τη συνάδελφο από την Ουγγαρία σε ό,τι αφορά τη χιλιομετρική αποζημίωση μόνο η άμεση, πιο άμεση ε, διαδρομή ε, μετράει ανεξάρτητα από το πώς ε, πήγες, από πού πέρασες, υπολογίζεται πιο άμεση διαδρομή, η χιλιομετρική. Υπάρχει ένα σύστημα που μετράει το κόστος ε, και ασφάλισης και τη, από τροχαίο ή από ατύγη βλάβη, το κόστος συντήρησης, όλα αυτά τα υπολογίζει. Και εγώ νόμιζα ότι είναι πολλά, αλλά όταν τα είδα, δεν είναι και τόσα πολλά τελικά. Γιατί δεν πληρώνεις μόνο για ένα αυτοκίνητο, πληρώνεις την ασφάλεια και... Μια φορά είδα ότι 35 χιλιόμετρα μόνο μου υπολόγισαν γιατί είναι αυτή άμεση διαδρομή. Das, ähm, auch και μπορούν να γίνουν διάφορες, ε, ε, διάφορα τρίκ τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι δεν ενδιαφέρει τόσο τι θα έπρεπε να πληρώσεις, τι πληρώνεις, ε, έξτρα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι τι απόσταση υπολογίζεται, που είναι η πιο άμεση. Το θέμα να μην χάσουμε το μέτρο με τη, τα διοικητικά έξοδα, τι δαπάνες. Ja, äh, ό,τι αφορά την κυρία Τσε για τα αυτοκίνητα δεν ε, κυκλοφορούν άδεια τα υπηρεσιακά οχήματα αυτά. Παραδείγματο χάρη παιδιά που συνοδεύονται, μάλλον γονεί που συνοδεύονται παιδιά του, ή έγκυση Υπάρχουν κάποιοι κανόνε τέλο πάντων ε, μπορούν δηλαδή να συνοδεύονται, ε, μπορούν να πάρουν κάποιους ε, οι λιμουζίνες αυτές. Σίγουρα δεν έχει κανένα νόημα να κυκλοφορούν άδεια, αλλά υπάρχουν για συγκεκριμένες ομάδες κάποια πράγματα, κάποιες δυνατότητες. Ό,τι αφορά τη γενική αποζημίωση εξόδων στην προηγούμενη θητή, είχα κάνει μια πρόταση στο Προεδρείο σε ό,τι αφορά αυτή την αποζημίωση αποφάσισε να συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας ε, το Προεδρείο που συνεδρίαζε για 1,5 χρόνο και μετά επιλέξαν δύο επιλογές ε, και το ε, Προεδρείο χρειάστηκε μετά από αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων μελών του Προεδρείου να ψηφίσει και ψηφίστηκαν αυτοί οι νέοι κανόνες τελικά εγώ και από την εμπειρία μου είμαι ότι θα συνεχίσει να απασχολεί και τον Ιν Προεδρείο Υποζημίωση Γενικών Εξόδων. Δεν ξέρω αν θα συγκροτηθεί η ομάδα εργασία ή θα τον λάβει κάποιον πρόεδρο, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα με εξέπληξε ιδιαίτερα αν ε, δεν ξανάνοιγε το ζήτημα αυτό και ίσως να ήδη να συζητείτε και θα συζητηθεί ίσως και στις αρχές Οκτωβρίου τώρα. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει τώρα αυτή η δυνατότητα εθελοντικά να υπάρχει αυτό το νομοθετικό footprint, ε, αποτύπωμα για τους ηγητές κτλ. Αυτό γίνεται στην αρχή Είμαστε στην αρχή μάλλον και δεν ε, έχουμε ακόμη πολλές συζητήσεις, δεν ε, έχει ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία πλήρως, αλλά μπορούμε να ενημερώσουμε τους ε, βουλευτές αν θέλετε και κάποια στιγμή στη θητεία, στη διάρκεια της θητείας θα μπορούσαμε να δούμε πώς οι βουλευτές το χρησιμοποιούν αυτό σε σχέση με το σύνολο των λεφτών. Κυρία Χολμάιερ, νομίζω απάντησε ήδη ε, το θέμα των ε, μετακινήσεων ε, εντό των κρατών. Γιατί, ναι, γιατί με έχει απασχολήσει εμένα προσωπικά το θέμα, κυρία Χολμάιερ. Υπάρχουν για πολλά άλλα και γι' αυτό λοιπόν κανόνες που έχουν, έχει επεξεργαστεί το Προεδρείο. Αν θεωρήσει το Προεδρείο ότι χρειάζεται να διορθωθούν, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα υπάρξει μια επεξεργασία των ε, διατάξεων υπάρχουν ε, ενδεχομένως ε, θέματα που δεν είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των όλων των μελών και υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους ό,τι αφορά τα νέα γραφεία και τις παροχές σε ό,τι αφορά την διευθύντρια του τμήματος που είναι και εδώ είναι η κυρία Κάρτιν και Άρμιν ε, καλό είναι να λέμε τα ονόματα για να είναι γνωστά και δούλεψαν μάλιστα αυτοί και το καλοκαίρι πολύ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής ε, των οδηγών για τους βουλευτές θα δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να είμαστε πιο ευέλικτοι. Ε, εξαρτάται και από το αν περιμένει και κάποιος άλλος με στο αυτοκίνητο το πρωί το βράδυ, αλλά θα το ξαναδούμε. Και σίγουρα με το νέο σύστημα πληροφορικής θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση και τον Νοέμβριο θα δούμε αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ερώτηση της κυρίας Χολμάιερ. Υπάρχουν χώρες που δεν προβλέπουν καν ε, κανονική σύνταξη για τους βουλευτές, Ιταλία, Γαλλία αλλά ε, αυτό ε, το υποκαθιστά η ε, πρόβλεψη από, τη, από τον νησιακό προπολογισμό που δίνει χρήματα. Δηλαδή όταν δεν μπορεί να παίρνει εθνική σύνταξη αυτός ο βουλευτής υπάρχει η δυνατότητα ιδιωτική σύνταξη. Υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλιο για τους Ταλούς και Γάλλους βουλευτές που εξασφαλίζει τη σύνταξη αυτούς που δεν θα έπαιρναν στην Ιταλία στην Γαλλία, επαναλαμβάνω, εθνική σύνταξη. Θα μπορούσαν βέβαια να γίνουν μέλη του Επικουρικού Συνταξιδοτικού Ταμείου Γάλλοι και οι Ιταλοί Ευρωβουλευτέ για να πάρουν την πρόσθετη σύνταξη. Άρα, όλοι οι βουλευτέ παίρνουν σύνταξη από το Εθνικό Συνταξιδοτικό Σύστημα είτε για του Ιταλού και του Γάλλου, μέσω ε, σχετική από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά μπορεί να ε, έχει δικαίωμα σε επικουρική σύνταξη οποιοδήποτε βουλευτή από το Συνταξιδοτικό Ταμείο. Τώρα, τι θα πει αναλογική σύνταξη, σε ό,τι το ύψο τη σύνταξη μεταξύ των κρατών μελών, οι διαφορέ ήταν δραματικέ. Υπήρχαν βουλευτέ που έπαιρναν μια πάρα πολύ χαμηλή σύνταξη και άλλοι που πέραν μια πάρα πολύ υψηλή σύνταξη. Τώρα με το καταστατικό το πρόβλημα αυτό ρυθμίστηκε, αλλά υπάρχουν τέτοιες ε, περιπτώσεις. Μετά από πολλά πολλά χρόνια βουλευτικής ε, δραστηριότητα να παίρνουν ε, κάποιοι πολύ λίγοι σύνταξη. Οπότε αυτή η δική σύνταξη, η επικουρική σύνταξη προσλαμβάνει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη τελικά αυτή που τους προσφέρεται μέσω του επικουρικού αυτού ταμείου από αυτή που παίρνουν στη χώρα τους. Πολύ ωραία. Αυτές ε, ήταν λοιπόν οι ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ο κύριος Κούς έχει άλλη μία ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να λάβω το λόγο. Το ζήτησα και προηγουμένως, δεν με είδατε κάπως. Συγγνώμη, συγγνώμη που δεν σας είδα. Λοιπόν, να κάνω μία ερώτηση. Επειδή εδώ ε, ρωτήθηκαν τα πάντα, κατ' ουσίαν δεν ρωτήθηκε κάτι συγκεκριμένο πρέπει να πω αυτό με εξέπληξε λιγάκι και γι' αυτό και εγώ να κάνω κάποιες έτσι ερωτήσεις. Και εγώ είμαι καινούριο. Βεβαίως ε, διάβασα το κόκκινο βιβλιαράκι για τα δικαιώματα των βουλευτών ε, και κάπου νομίζω διάβασα ότι η αποζημίωση, η μερίσια αποζημίωση καταβάλλεται μόνο αν είναι κανείς παρόν τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα. Ισχύει αυτό και πώς το ελέγχεται. Γιατί όταν μπαίνω στο κοινοβούλιο, πράγματι χρησιμοποιώ ε, το μπάτς μου. Ε, για να βγω όμως δεν χρειάζεται. Μπαίνω και βγαίνω μάλλον έτσι. Ε, γιατί οι κυλιόμενες πόρτες ε, μου επιτρέπουν να βγω χωρίς να πατήσω τίποτα. Και ερωτώ. Εμείς οι βουλευτές ε, καταγράφεται το τι κάνουμε, πότε μπαίνουμε και πότε βγαίνουμε με αυτό το γενικό σύστημα καταγραφής. Ε, γιατί έτσι μπορεί κανείς να αποδείξει πότε μπήκε και πότε βγήκε. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω αφορά το ταξίδι. Βρυξέλλες, Στρασβούργο ή οτιδήποτε. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ευρωβουλευτή ε, που ζει κάπου κοντά ή ας το πούμε και αλλιώ. Ε, αν πάρει κανείς καθοδόν κάποιον στο αυτοκίνητο και συνεχίσουν μαζί, ο ένας θα πάρει κάτι, ο άλλος δεν θα πάρει τίποτα. Κοιτάξτε, ε, με το δικό μας το εθνικό σύστημα, αν κάποιος χρησιμοποιεί δημόσιο αυτοκίνητο και πάρει και άλλον συνεπιβάτη, θα επιβραβευτεί. Δεν θυμάμαι, νομίζω είναι 3 σέντ το χιλιόμετρο, κάτι τέτοιο. Ε, γιατί δεν το σκέφτεστε κι εσείς αυτό. Έτσι μπορεί να μειωθεί το κόστος. Το να κάνουν δύο διαφορετική εκαθάριση ε, είναι πολύ πιο ακριβό από το να πάρει κανείς ένα πριμ επειδή πήρε συνεπιβάτη. Ε, έχουμε τους, τους νέους χώρους που μας δώσατε, πάρα πολύ ωραίοι χώροι αυτοί. Ε, και εκεί υπάρχουν αυτό που είπαμε σαλονάκι. Δηλαδή εκεί είναι δύο πολυτρόνες και ένα στρογγυλό τραπέζι από πέτρα. Και άκουσα ότι αυτά τα τραπεζάκια είναι πολύ ακριβά. Ε, μάλλον οι πολυθρόνε είναι πολύ ακριβές. Κόστησε κάθε μία από αυτές 1.600 ε, ευρώ, γιατί αν είναι 1.600 ευρώ, τότε θα μας κριτικάρουν ε, πάλι, θα μας επικρίνει η κοινή γνώμη. Κοιτάξτε, λέει η πρόεδρος, μην τα λέτε αυτά, γιατί ξέρετε κάτι, ε, κάπου το διαβάσει, κάποιο το είπε, δεν ισχύει, θα το διαψεύσει το κοινοβούλιο, αλλά μεταξύ τι γίνεται, μένει λάσπη. Δηλαδή όλοι θα διαβάσουν ότι κόστησε η πολυθρόνα 1600 ευρώ και κανείς δεν θα διαβάσει τη διάψευση. Σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος, μην ρωτάτε τώρα οτιδήποτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτάτε θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας, την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. the I would just like to quickly follow up. Να συνεχίσω λίγο για τα αυτοκίνητα για το Στρασβούργο. Τα αυτοκίνητα μπορεί να μην είναι εντελώς άδεια, αλλά είμαι βεβαία ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαθέσιμη χωρητικότητα. Παρακαλώ να το εξετάσετε να δείξετε το ενδιαφέρον σας, να δείξει και ο κόσμος την δυνατότητα. Δεν είναι πολιτικό, θα γλιτώσει πολλά χρήματα και θα βοηθήσει πολλούς να ταξιδέψουν με αξιοπρέπεια. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και απρόβλεπτη, πολύ απρόβλεπτη. Αυτό μου γέννησε μία ιδέα και μιας και μου είναι λίγο σπάνιο θα σας την μεταφέρω. Νομίζω ότι οι κοσμήτορες θα μπορούσαν να οργανώσουν μία συνάντηση υποδοχής των βουλευτών για να απαντήσουν σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Τα δύο τρίτα είναι νέοι βουλευτές. Οπότε ένας κοσμήτορας και ένας εκπρόσωπος του γραφείου σας μία φορά την εβδομάδα να είναι σε θέση να απαντήσει στις πρακτικές ερωτήσεις μας. Και εγώ ξεκίνησα εδώ και δύο εβδομάδες και να πω ότι μία ερώτηση πάρα πολύ απλή πάντα είναι πιο περίπλοκη και σύνθετη. Αυτό το οποίο θεωρείται αυτονόητο μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να λύσει κανείς. Παίρνω το παράδειγμα των παιδικών σταθμών. Ε, όλοι συμπαθούμε ε, ε, μάλλον μας αρέσει η ιδέα ότι πρέπει οι βουλευτές να πηγαίνουν το παιδί του στον παιδικό σταθμό το πρωί. Όταν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνει μια, θα έλεγα, παράκαμψη μισή ώρα, τώρα είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να το κάνει αυτό. Λοιπόν, είναι μια απλή ερώτηση μια περίπλοκη απάντηση. Αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα σε αυτούς που κατοικούν στις Βρυξέλλες και αυτούς που είναι εκτός Βρυξελών. Γιατί για να έχουμε το παιδί μας σε παιδικό σταθμό σημαίνει ότι μένουμε μόνιμα εδώ. Πώς αντιμετωπίζουμε τη διαφορά εδώ, την αποδεχόμαστε ή όχι. Ένας κανόνας ο οποίος φαίνεται λογικός και προκαλεί συμπάθεια, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία είναι περίπλοκη. Να Ένα παράδειγμα λοιπόν των θεμάτων τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν σε επίπεδο κοσμητόρων με την πολύτιμη βοήθεια του Γενικού Γραμματέως. Τέλεια η ιδέα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στο Γενικό Γραμματέα. Και εγώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας, γιατί πράγματι πολλά από τα θέματα που έτσι είναι θέματα που αφορούν τους κοσμήτωρες. παρόλα όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Ε, κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε συστηματικό έλεγχο ευρωβουλευτών με το σύστημα καταγραφής και σε τελική ανάλυση δεν θα βοηθούσε κάτι τέτοιο, γιατί οι ευρωβουλευτές ε, κάνουν δουλειά όχι μόνο εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και εκτός Κοινοβουλίου. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους ε, συνεργάτες, ε, έχουμε ένα σύστημα για συνεπιβάτες Δηλαδή, ας πούμε ότι ένας υπάλληλος μας πάει σε αποστολή ε, και πάρει και κάποιον άλλον μαζί του, ε, τότε ο ε, οδηγός επιβραβεύεται γιατί χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του και έκανε εξοικονόμηση χρημάτων. Τώρα, τα έπιπλα για τους ευρωβουλευτές τα πήραμε με leasing αυτή τη φορά, που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, να προσαρμόσουμε τα έπιπλα στις ανάγκες των βουλευτών. Ε, γιατί ο ένας θέλει μεγάλο τραπέζι, ο άλλος μικρό, ο άλλος θέλει πολυθρόνες. Ε, όταν είναι κάτι λογικό, από τον Νοέμβρη θα μπορεί κάθε ευρωβουλευτής να διαλέξει μόνος του τα επιπλά του. Και σας είπα, δεν θα τα αγοράσουμε, θα τα εκμισθώσουμε με το σύστημα του leasing τα έπιπλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ε, παλαιότερα, ξέρετε τι γινότανε, τα έπιπλα που αγοράζαμε, τελικά ε, τα πετάγαμε, είχαμε ένα ολόκληρο νεκροταφείο παλιών επίπλων. Αυτό το σύστημα με το leasing είναι τέλειο. Ε, γιατί με τους καινούριου, οι καινούργοι δεν ήθελαν κάτι που είχε ένας παλιός, πηγαίναν όλα στο υπόγειο, ε, τώρα το βρίσκω πολύ καλό ότι υπάρχει προσαρμογή στις ανάγκες, γιατί ο κάθε βουλευτής έχει τις δικές του ανάγκες. Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Γραμματέα που πραγματικά απάντησε σε πληθώρα ερωτήσεων ε, και ευχαριστούμε και για την ιδέα που εξέφρασε ο Κοσμήτορας. Ευχαριστώ όλους ε, τους αδέλφους. Αύριο το πρωί θα συναντηθούν οι συντονιστές Γεια σας, καλό βράδυ.